Ladies and gentlemen, good afternoon. Please be seated. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καθίστε παρακαλώ. Όπως είπαμε νωρίτερα, θα αρχίσουμε την απογευματινή μας συνεδρίαση με ένα εργαστήρι, ένα workshop που αφορά την ρωσική στρατιωτική παρουσία στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης παρακαλώ βάλτε τα ακουστικά σας γιατί θα μιλήσω και πολωνικά. Ε, έχουμε μιλητές λοιπόν για το θέμα αυτό το τόσο ενδιαφέρον. Καταρχάς έχουμε έναν αναλυτή από ένα πολωνικό think tank TISM Άννα Μαρία Τίνερ που εδώ και πολλά χρόνια ασχολείται με αυτό το θέμα θα είναι ο πρώτος μας ομιλητής για αυτό το ζήτημα. Δεύτερος προσκεκλημένος και Μίνεσιαν, δημοσιογράφος Λεμόντ. που ασχολείται και πάλι πολλά χρόνια με την περιοχή αλλά μιας και έχουμε λίγο χρόνο στη διαθέσή μας και η μερίσια διάταξή μας είναι γεμάτη χωρίς να καθυστερήσουμε άλλο θα δώσω το λόγο στους ομιλητές έχετε το λόγο παρακαλώ Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε ευχαριστώ που μας δίνετε την ε, ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της έρευνάς μας για ζητήματα ασφάλειας στην μετασοβιετική εποχή. Θα ξεκινήσω τώρα την παρουσίασή μου γιατί γνωρίζω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Να ξεκινήσω από πού έχει προέλθει αυτή η ρωσική στρατιωτική παρουσία ε, στην περιοχή μας. Βεβαίως πρέπει να πάμε πίσω στην εποχή της Σοβιετικής Ένωσης και στο σύστημα ασφάλειας ε, της Σοβιετικής Ένωσης. Υπήρχαν τρεις ομόκεντρικοί κύκλοι, ας πούμε. Ε, υπήρχαν τα κράτη δορυφόρη της ε, ε, Σοβιετικής Ένωσης, ε, Τσεχοσλοβακία, Πολωνία και χώρες οι οποίες ήταν υπό την άμεση ετοιμότητα. Κάντε. Δεύτερος και ομόκληρος κύκλος ήταν τα κράτη των Βαλκανίων, η Ουκρανία ή η Λευκορωσία. Εκεί υπήρχαν στρατιωτικές βάσεις και στρατεύματα του Σοβιετικού στρατού. Τα στρατεύματα αυτά δεν είχαν πλήρη ετοιμότητα, αλλά ήταν εξοπλισμένα και ήταν σε ένα μέσο επίπεδο ετοιμότητας. Και ένα, ένας τρίτος ε, ομόκεντρος κύκλο ήταν αυτός εντός της Σοβιετικής επικράτειας που ήταν ε, και στο χαμηλότερο επίπεδο ετοιμότητας. Έτσι λοιπόν έχει προκύψει η ρωσική στρατιωτική παρουσία σε χώρες όπως η Λευκορωσία και η Μολδαβία σήμερα. Όσον αφορά τη Λευκορωσία υπάρχουν μια σειρά από έγγραφα βάσει των οποίο η Λευκορωσία και η Ρωσία συνεργάζονται σε θέματα άμυνας. Τα πιο σημαντικά έγγραφα, τέσσερα τον αριθμό είναι, το πρώτο έγγραφο αποτελεί μια συμφωνία σύνδεσης. Δεύτερο είναι ε, η συμφωνία για την διαφύλαξη των εξωτερικών συνόρων των χωρών και την δημιουργία κοινών αμυντικών στρατευμάτων. Τρίτον είναι η αμυντική συνεργασία μεταξύ Λευκορωσίας και Ρωσίας. Και τέταρτο στοιχείο είναι δύο έγγραφα που αφορούν την στρατιωτική υποδομή, την ρωσική στρατιωτική υποδομή, στο έδαφος της Λευκορωσίας. Γιατί είναι σημαντική η Λευκορωσία ε, για τη Ρωσία. Κοιτάξτε το χάρτη. Τα σύνορα Ε, έχουν μετακινηθεί κατά 540 χιλιόμετρα και επίσης βρίσκεται πολύ κοντά η χώρα αυτή στην Μόσχα. Οι δύο χώρες λοιπόν έχουν συνάψει συμφωνία ε, για συνεργασία σε ζητήματα ασφάλειας. Όσον αφορά τη σημαντικότερη στρατιωτική υποδομή στην ε, Λευκορωσία, πρόκειται για τους σταθμούς στο Παλεβίτσε, ένα σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας της ε, Ρωσίας και υπάρχουν και διάφορες άλλες εγκαταστάσεις για την ε, επικοινωνία με ρωσικά υποβρύχια. Εδώ στο χάρτη βλέπετε την, ε, το σημείο στο οποίο είναι η βάση. Εδώ είναι η βάση. Εδώ βλέπετε το Χανσεβίτσα στην, στην, στον, στην νότια Λευκορωσία η Ρωσία δεν έχει εγκαταλείψει καμία από τις δύο ε, στρατιωτικές βάσεις. Θα τις διατηρήσουν έως το 2020 σίγουρα και θα κοιτάξουν να επεκτείνουν τη λειτουργία τους και για, το, για την περίοδο μετά. Τώρα, για τις επιχειρήσεις των δύο χωρών υπάρχουν δύο κατηγορίες βασικές. Πρόκειται για τις ε, δυτικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις ασπίδας. Η τελευταία έγινε το 2013 με σενάριο βάσει του οποίου Λευκορώσοι και Ρώσοι ασκούνταν σε συνθήκες γεγονότων όπως αυτά που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης. 70 τάγκς πήραν ε, μέρος σε αυτή την άσκηση, 60 ελικόπτερα, συστήματα πυράβλων, αλλά και πολεμικά σκάφη, γιατί η άσκηση αυτή συμπεριέλαβε και χώρες της, και τη Βαλτική θάλασσα. Όσον αφορά την ασπίδα, η τελευταία σχετική άσκηση έγινε το Σεπτέμβριο του 2015 και η ελιγμή αυτή, η άσκηση αυτή, συμπεριέλαβε, στην άσκηση αυτή συμμετείχαν 7.000 Ρώσοι στρατιώτες και 1.000 Λευκορώσοι στρατιώτες με 100 τάγκς και 85 μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα. Η άσκηση έγινε στο μεγαλύτερο μέρος της στο Λένιγκρατ και στο Καλίνιγκρατ. Αυτές, αυτοί οι αεροπορικοί ελιγμοί χρησιμοποιούνται κυρίως από τη Λευκορωσία για να διατηρείται το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και είναι αξιοσημείωτο επίσης το γεγονός ότι τα ρωσικά στρατεύματα όχι τα λευκορωσικά στρατεύοντα, με συγχωρείτε, λαμβάνουν εντολές στα ρωσικά, εκπαιδεύονται στα ρωσικά, στη, στη ρωσική γλώσσα δηλαδή. Θα μπορούσε να πει κανείς δηλαδή ότι λόγω της συμφωνίας σύνδεσης και του κοινού εναέριου χώρη, οι Ρώσοι με πολύ μεγάλη ευκολία ε, ελέγχουν την επικράτεια της Λευκορωσίας. Να περάσουμε τώρα στη Μολδαβία. Εδώ η κατάσταση είναι η εξής. Μιλάμε για την υπερδνηστερία, μια αποσχιστική δημοκρατία που δεν αναγνωρίζεται από, κανένα, από, κανένα, από κανένα κράτος. Τα πράγματα ξεκίνησαν το 1990 και την τότε κατάσταση στην ε, πρώην Σοβιετική Ένωση, όπου υπήρχαν διάφορες τάσεις αποσχιστικές και εθνικιστικές σε διάφορες περιοχές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Σε εκείνη τη φάση λοιπόν η μειονότητα της υπερνηστερίας κήρυξε την ανεξαρτησία της. Οι σειράξεις ξεκίνησαν το 1991 και για να διατηρηθεί η η ανεξαρτησία κομβικό ρόλο έπαιξε το 14ο τάγμα υπό τον ε, στρατάρχη Λέμπιετς. Το 1994 υπεγράφει ανακοχή και έκτοτε στην Μολδαβία υπάρχουν στρατεύματα εδάφους. Αποκαλούνται στο μεγαλύτερο βαθμό τους, ε, στο μεγαλύτερο μέρος τους ως ειρηνευτικές δυνάμεις, συμπεριλαμβάνουν Ρώσους και υπάρχει, υπάρχει και ένας μικρός αριθμός στρατιωτών που φυλάσσουν τις παλιές στρατιωτικές αποθήκες που υπάρχουν εκεί από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης. Μέχρι στιγμής δεν έχει εξευρεθεί μια καλή λύση και εδώ βλέπετε στο, στη διαφάνεια τις στρατιωτικές αποθήκες των Ρώσων και την υπερμηνιστερία. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι η εξής. Επειδή η Ουκρανία έχει αρνηθεί το δικαίωμα διέλευσης ε, σε ρωσικά στρατεύματα. Οι Ρώσοι στρατολογούν ανθρώπους από τον τοπικό πληθυσμό ρωσικής καταγωγής και επηρεάζουν και την σύνθεση των στρατευμάτων που ε, βρίσκονται ε, στην συγκεκριμένη περιοχή. Συνολική δύναμη των στρατευμάτων ανέρχεται σε 1.500 άτομα και σε αυτά προστίθενται και άλλοι 400 στρατιώτες που φυλάσσουν τις στρατιωτικές αποθήκες. Ε, κάνουν ασκήσεις ε, και μια δυσκολία που υπάρχει για την ε, Μολδαβία και στην επικοινωνία της με την Ουκρανία είναι ότι υπήρξε το 2014 μια απειλή λόγω πιθανής διέλευσης στρατευμάτων μέσω υπερδενιστερίας προς την Ουκρανία. Τώρα, για να περάσουμε και στην περίπτωση της Ουκρανίας. Πριν από το 2014, η Ρωσία και η Ουκρανία ε, είχαν ε, πολλές συμφωνίες μεταξύ τους, όπως η Συμφωνία Φιλικών Σχέσεων μεταξύ των δύο χώρων, που ακυρώθηκε από το Ουκρανικό που επρόκειτο μάλλον να ακυρωθεί από το Ουκρανικό Κοινοβούλιο, αλλά η διαδικασία έχει κολλήσει. Επίση υπήρχε συμφωνία στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και συμφωνία για την ε, παρουσία ε, ναυτικού, πολεμικού ναυτικού στη σεβαστόπολη στην Κρυμαία. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι το Ρωσικό Κοινοβούλιο έχει αποσυρθεί από αυτή την συμφωνία ενώ οι Ουκρανοί δεν έχουν καταφέρει να το κάνουν ακόμα. Και ε, το 2014 μετά την επανάσταση της αξιοπρέπειας τα πράγματα άλλαξαν οπότε και οι Ρώσοι με βάση τη συμφωνία για τη Μαύρη Θάλασσα, για το στόλο στη Μαύρη Θάλασσα, αποφάσισαν να αυξήσουν τα στρατεύματα εδάφους και αναφέρεται ότι αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας υπάρχουν 24.000 στρατιώτες Ρώσοι, οι οποίοι έχουν ενισχύσει το σύστημα προστασίας της, ε, των ακτών, ε, διαθέτουν πολεμικά αεροσκάφη, μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, τα οποία μπορούν να πολεμήσουν και με πολεμικά σκάφη και με βάση το ρωσικό δόγμα εξετάζεται και το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων καθώς εξετάζεται και το ενδεχόμενο να επανατοποθετηθούν σε άλλα σημεία ε, πυρηνικές κεφαλές. Η Ρωσία λοιπόν έχει ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της στην περιοχή. Τώρα, για τον Ντομπάς και την περιοχή του Ντονιέτσκ, εκτιμάται ότι οι Ρώσοι έχουν 7.000 στρατιώτες ξηράς αυτή τη στιγμή. Και τα στρατεύματα αυτά, κατά κύριο λόγο, ελέγχουν την περιοχή. Τώρα, τι είδους εξοπλισμός υπάρχει στην περιοχή του Ντονιέτσκ. Εκτιμώ ότι υπάρχουν 100 περίπου οπλικά συστήματα, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, ε, γιατί υπήρχε πριν από τις εξελίξεις των τελευταίων ετών ε, και ε, ουκρανικός εξοπλισμός εκεί. Επίσης, τα σύνορα, ε, τα ουκρανο-ρωσικά σύνορα δεν ελέγχονται από την Ουκρανία, οπότε η Ρωσία μπορεί να μεταφέρει στην περιοχή αυτή όσο εξοπλισμό θέλει χωρίς να την ελέγχει κανείς. Επισήμω, ε, θεωρητικά, σύμφωνα με, τη με του, Προέδρου Πούτιν, δεν υπάρχουν στρατεύματα ξηράς. Επίσης, βλέπουμε ότι οι Ρώσοι έχουν ενισχύσει την παρουσία τους στα ρωσικά ε, σύνορα με την Ουκρανία και με την Λευκορωσία και σύντομα, πρόσφατα αποφάσισαν να δημιουργήσουν τρία νέα τάγματα τα οποία ε, θα ε, έλεγχαν τα σύνορα με την Ουκρανία και με την Λευκορωσία. Συμπερασματικά, όσον αφορά την ρωσική παρουσία σε συγκεκριμένες χώρες, στην Λευκορωσία έχουν 600 στρατιώτες ξηράς. Πρόκειται για τους ανθρώπους που συντηρούν τις δύο στρατιωτικές βάσεις που υπάρχουν στη χώρα. Στην Μολδαβία υπάρχουν περίπου 1.500 στρατιώτες των ηρωνευτικών δυνάμεων και άλλοι 400 που φυλάσσουν τις στρατιωτικές αποθήκες. Στην Ουκρανία υπάρχουν περίπου 24.000 στρατιώτες στην Κρυμαία και άλλοι 7.000 στο Ντομπάς. Τα στοιχεία μπορείτε να τα βρείτε και στο έγγραφο που έχουμε προετοιμάσει για εσάς, για την σημερινή συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και αν έχετε ερωτήσεις θα είμαι στη διάθεσή σας φυσικά. Επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο στον κύριο Γκάιτ Μενετσιάν από τη Λεμόν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι είμαι ερευνητή για στρατηγικές έρευνες και δεν εκπροσωπώ την εφημερίδα Le Monde. Μου φαίνεται ότι είναι χρήσιμο να κάνω αυτή τη διευκρίνηση. Κανένα πρόβλημα κύριε Πρόεδρε. Αυτό που θα ήθελα να πω καταρχάς πέρα από το έγγραφο που λάβατε σχετικά με τις λεπτομέρειες της ρωσικής παρουσίας στο Νότιο Κάφκασο, θα ήθελα να βγάλουμε ορισμένα συμπεράσματα σε ό,τι αφορά την παρουσία των Ρώσων στο Νότιο Κάφκασο. Έξι πράγματα, έξι διδάγματα. Το πρώτο είναι συγκυριακό. Από τον πόλεμο του 2008 μεταξύ της Ρωσίας και της Γεωργίας καταγράφεται μία ενίσχυση της ρωσικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή. Η Ρωσία ακολουθεί μία διαδικασία εναρμόνισης και μία πολιτική στρατιωτικής συνοχής. Οι, συμφωνίες που έχουν υπογραφεί μεταξύ Ρωσίας, Αυγαζίας και Ρωσίας και Αρμενίας είναι σχεδόν η ίδια, σχεδόν ταυτόσιμες προ προς το περιεχόμενό τους. Αυτή η διαδικασία ολοκλήρωσης θα συνεχιστεί και στο μέλλον θα λέγαμε. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το στρατηγείο των στρατηγικών δυνάμεων των ρωσικών στρατευμάτων στην Απγαζία και στην Αρμενία βρίσκεται στο μπροστό. Δεύτερο. Το δεύτερο δίδαγμα είναι ιστορικού χαρακτήρα. Στην, στο Νότιο Κάφκασο η Ρουσία προωθεί μια εικόνα σοβιετική και αυτοκριταρική, προσπαθεί να ενσωματώσει τόση αυτή την περιοχή την εποχή των Τσάρων, η κατάκτηση ήταν πρωτίστως στρατιωτικού χαρακτήρα, μακρά και αιματηρή πριν να γίνει πολιτιστική. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, τελείωσε το 21, ο κόκκινος στρατός συμπεριέλαβε με την βία την, ε, το Κάφκασο. Σήμερα ακόμα και αν ο πρόεδρος ο Πούτιν εκφράζει την αντίθεσή του στη ε, ε, Μόσχα. Υπάρχει η επιθυμία να εσωματωθεί και πάλι αυτό στα πλαίσια ενός πολυπολικού κόσμου όπου η Ρωσία θα ήταν ένας πόλος ε, έλξης. Με λίγα λόγια, η Ρωσία γνωρίζει μόνο τη λογική της ισχύω προκειμένου να σκίσει την εξουσία της. Το τρίτο μάθημα που μάθαμε από τη ρωσική παρουσία, τη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, προκύπτει από το δεύτερο δίδαγμα και είναι στρατηγικής ε, υφής. Η διαδικασία αυτή επανόδου της περιφερειακής επιρροής ασκείται με διαφορετικό τρόπο σε τακτικό επίπεδο. Πράγματι, η Ρωσία δεν υιοθετεί την ίδια διαδικασία σε ό,τι αφορά τις τρεις δημοκρατίες και για το λόγο αυτό μπορούμε να μιλήσουμε τον κανόνα των τριών σε. Κοπερασιόν, συνεργασία με την Αρμενία, το Γερεβάν και το, το μόνο νότια της Κορέας, η Μόσκα και το Γερεβάν έχουν παράλληλα συμφέροντα στην περιοχή, μπροστά στην ιστορία και την απειλή της Τουρκίας στην περιοχή. Η Ρωσία πάντοτε θεώρησε τα σύνορα με την Τουρκία σαν μια πηγή κινδύνου, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα. Εξ της ασφάλειας των Αρμενίων που έχουν πληγεί από τη γενοκτονία την οποία αρνούνται οι Ρώσοι, το Γερβάν βλέπει μια πραγματική απειλή. Η Τουρκία μόνο μερός έχει κλείσει τα σύνορά της με το Γερβάν το 1993 ως ένδειξη ελληνικής με τον Πακού, το οποίο ιτήθηκε από τους Αρμένιους στον πόλεμο του Ναγκόρ Καρμπάκ. Δεύτερο, σε, μετά την κοοπερασιόν, συνεργασία, κομφροντασιόν, αντιπαράθεση με τη Γεωργία. Η Ρωσία θέλει να α, μην υπάρξει πλέον καμία ελπίδα ένταξη στην Ατλαντική Σημασία. Χρησιμοποιούνται διάφορα μέσα ως τρόπος πίεσης επί των Γεωργιανών. Τρίτο σε, κομφιζιόν, σύγχυση με το Αζερβαϊτζάν. Η Ρωσία δεν έχει πλέον στρατιωτικές δυνάμει στο Αζερβαϊτζάν μετά το, την, το κλείσιμο του σταθμού τη Γαμπάλα. Οι διμερεί σχέσεις Μπακού, Μόσχα είναι καλές, Εξαίρετε, θα λέγαμε. Γνωρίζουμε εδώ και μερικά χρόνια ότι η Ρωσία πούλησε για 4 ή 5 δολάρια εξοπλισμού, ε, στρατιωτικού εξοπλισμού στο Αζερβαϊτζάν παρόλη παρόλο το ότι είναι σε αυτές οι σχέσεις, παραμένει μια αμοιβαία υποψία. Το Μπακού φοβάται τη Ρώσο-Αρμενική Συμμαχία και κατηγόρησε τους Ρώσους ότι βοήθησαν τους Αρμένιους κατά τη διάρκεια του πολέμου του Καραμπάκ. Για τον Μπακού η Μόσχα είναι η υπέρ των Αρμενίων όταν η Ρωσία είναι αδύνατη και υπέρ του Αζερβαϊτζάν όταν η Ρωσία είναι ισχυρή. Από την δική της πλευρά η Μόσχα ε, είναι καχύποπτη για το Αζερβαϊτζάν, το οποίο δίνει προτεραιότητα στι σχέσει με την Τουρκία. Και στη Μόσχα θεωρείται ότι το Μπακού είναι υπέρ τη Ρωσία όποτε μπορεί και υπέρ τη ε, Τουρκία όταν πρέπει. Το τέταρτο μάθημα είναι τεχνικό και στρατιωτικό ε, στρατεύματα κατοχής ε, ε, και οι ε, ρωσικές δυνάμεις ακούν σχεδόν τους ίδιους εξοπλισμούς στις διάφορες βάσεις. Στην ουσία πρόκειται για στρατό ξηράς με άρματα μάχης και αυτό μας δείχνει ότι η χρήση τους είναι κατά αποκλειστικότητα τοπική. Παράλληλα υπάρχει διάθεση ενίσχυσης των οπλικών συστημάτων στις παράκτιες περιοχές της Μαύρης Θάλασσας με μια παρουσία στην Κρυμαία και στην Αυγασία σαν ένα είδος γεωγραφικής συνέχισης τη οποία τη σημασία δεν πρέπει να υποτιμάμε. Η άλλη τεχνική και στρατιωτική πτυχή έχει σχέση με την άλλη ισοτροφοδοσία. Για την ώρα, η βάση του τα μπροστά στην Τουρκία, στην Αρμερία ε, εφοδιάζεται ε, με νέριες μεταφορές από το Ιράν. Πράγματι, η Ρωσία ανοίγει τους σιδηροδρόμους μεταξύ της Αυγαζίας, της Γεωργίας και της Αρμενίας προκειμένου να σταλούν, να διακινηθούν ε, ε υλικά και άνθρωποι. Αυτό απαιτεί την βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας. Το πέμπτο μάθημα που έχουμε μάθει είναι παγκόσμιο χαρακτήρα. Η, Μόσχος, η Μόσχα κινείται σε ένα πολυπολικό κόσμο, όπου η Μόσχα θα προσπαθούσε να έχει μια ζώνη επιρροής. Εξ ονόματος αυτού του κόσμου η Αρμενία και η Ρωσία διαπραγματεύονται τη δημιουργία ενός συστήματος εναέριας κοινή άμυνας, όπως η Λευκορωσία και η Ρωσία στην Ευρώπη και ε, όπως γίνεται στην κεντρική ε, Ασία. Η Ρωσία έχει σκοπό να κινηθεί σε δύο χρόνους. Καταρχάς οι τρεις περιφερειακές συμφωνίες, μετά μία εναρμόνιση προκειμένου το σύνολο αυτών των στρατηγικών χώρων να είναι κάτω από την ίδια ομπρέλα, δηλαδή κάτω από τους Ρώσους. Ο πόλεμο στη Συρία προσδίδει μια παγκόσμια διάσταση στην ρωσική παρουσία στον Κάφκασο. Ακόμα και αν τα πράγματα δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί, το γεγονός ότι η Ρωσία ε, κινήθηκε προς τη Συρία ε, έχοντας ως ορμητήριο την Κασπία μας δείχνει ότι την περιοχή αυτή την αφορά η, η τρομοκρατία των τζιχαντιστών, μόνο ότι υπάρχει στην περιοχή ο Κάφκασος. Φάνηκε ότι διάφορες ρωσικές βάσεις που βρίσκονται στο νότιο Κάφκασο αυτή τη κυμερή είναι εκείνες που έχουν άμεση σχέση σε περίπτωση σύγκρουση με τη Συρία λόγω της γειτνίας με την Τουρκία η οποία είναι αντίπαλος της Ρωσίας στη Συρία και υπάρχει βεβαίω υπάρχουν αεροπορικές δυνάμεις στην αεροπορική βάση κοντά στο Γερεβάνο. Σε περίπτωση που η Ρωσία πάρει μέρο σε μία ενδεχόμενη ε, στο Ιράν, η, ε, το, το, ο, ο βασικός στόχος θα είναι το κυβερνή στην Αρμενία. Το τελευταίο πράγμα που θα μπορούσαμε να μάθουμε είναι τοπικού χαρακτήρα με τις συγκρούσεις. Λόγω των διαφορών με τη Γεωργία η Ρωσία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις της στην ε, Αμχασία. Σύμφωνα με τις ε, συμφωνίες που έχουν ε, υπογραφεί με τις δύο αυτές επαρχίες, οι οποίες αναγνωρίζονται ως ανεξάρτητα κράτη από τη Ρωσία. Στην ε, πλειοψηφία του Καραμπάκ η κατάσταση είναι κάπως διαφορετική. Η... Τότε με το άρθρο για την αμοιβαία βοήθεια σε περίπτωση εξωτερικής απειλής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά μόνο σε επίθεση κατά της Αρμενίας. Αυτό λοιπόν αποκλείεται αποκλεί το Καραμπάχ. Όπως είδαμε κατά τη διάρκεια του πολέμου των τεσσάρων ημερών, το 2016, τα σημεία βρίσκονται στα προσανατολά μεταξύ του Καραμπάκ και του Αζερβαϊτζάν και όχι όπως συμβαίνει παραβιάσεις της ε, πάψης ε, πυρός στα σύνορα μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερβαϊτζάν. Αυτό μας ε, κάνει να πιστέψουμε ότι το, το Μπακού χωρίς να έχει ξεκινήσει τις ε, ε, ενέργειες αυτές και όχι οι Αρμένοι οι οποίοι θέλουν να διατηρήσουν ε, την κατάσταση ως έχει. Παρόλα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη αυτό η Αρμενία διαπραγματεύεται μια στρατηγική συμφωνία σε περίπτωση επίθεσης. Αυτό σημαίνει ότι αυτόματα μια συμμετοχή της Αρμενίας σε αυτό τη σύγκρουση, ότι θα αυξηθεί ο κίνδυνος σύραξης, αλλά και ότι θα γίνει, θα αναγνωριστεί η ανεκκρατησία του Καραμπά. Όλα αυτά βεβαίως τώρα βρίσκονται στην τελική, στην τελική τους φάση. Ευχαριστώ, είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Uh, Ευχαριστώ. Πριν να δώσω το λόγο στους ομιλητές, βλέπω ότι ζητούν διαφορετικό λόγο. Θα ήθελα και εγώ το λόγο γι' αυτό το θέμα. Έχουμε και την παρέμβαση του κ. Μινεσιάν. Είναι πολύ δύσκολο για μένα ως πρόεδρος αυτής της επιτροπής αλλά και ως πολίτης Πολωνίδα βλέποντας όλη αυτή την εμπειρία, όλες αυτές τις χώρες, τα έθνη τα οποία συζητάμε πρέπει καταρχάς να πούμε ότι είναι χώρες κυρίαρχες και όχι παιχνιδάκια στα χέρια των Ρώσων. Γιατί βλέπουμε ότι αυτή είναι η λογική τους. Βέβαια, είναι θέμα συνένεσης και διεθνούς αναγνώρισης εδώ στο Κοινοβούλιο. Και ιδιαίτερα στην Επιτροπή μας, στην ΣΕΝΤΕ, είναι περισσότερο από προφανές ότι η Νότιο Οσετία και η Απχαζία αποτελούν ε, εδάφη υποκατοχή της Γεωργίας και ότι το Ναγκρόνο Καραμπάχ δεν είναι μια δημοκρατία. Επειδή άκουσα την αγγλική μετάφραση λέει πρόεδρος, οπότε δεν ξέρω ακριβώς εσείς πώς το μεταφέρατε. Αν υπήρξε δηλαδή κάποια παρερμηνία. αλλά εμείς αναμένουμε οι χώρες αυτές να είναι δαφικά ακέραιες. Αυτή είναι η δικιά μου η αντίληψη και νομίζω αυτό σχημάτισα από την παρουσίασή σας. Επειδή η χώρα η οποία οπωσδήποτε ωφελείται από το πρόσφατο ξέσπασμα τη σύραξη στον Αγκόνο Καραμπάχ, Αζερβαϊτζάν, Αρμενία και όχι μόνο εκεί, αλλά και σε άλλα εδάφη που κατέχει το Αζερβαϊτζάν. Η χώρα αυτή λοιπόν που ωφελείται, ξαναλέω, είναι η Ρωσία, η Ρωσική Ομοσπονδία. Καταρχάς, επειδή τους παρέχει ένα οικονομικό πλεονέκτημα σε εποχές ε, τιμών, χαμηλών τιμών ενέργειας μέσω της πώλησης των όπλων και βεβαίως εδώ έχουμε και ένα θέμα επιρροής. Εμείς δεν είμαστε τόσο βέβαιοι όσο εσείς για το, ποιο ξεκίνησε τη σύραξη αυτή και ποιος ωφελείται περισσότερο. Δεν είναι ακόμα α, ξεκάθαρο. ο Στρογεύσκη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κρίμα που έχουμε μόνο μια ώρα στη διάθεσή μας, λίγος ο χρόνος. Να ρωτήσω κάτι και τους δύο εισηγητές μας. Με την πρώτη συγκεκριμένα να ρωτήσω πρώτα. Η κρίση αυτή στην Κρυμαία φαίνεται ότι δεν μπορούσε να προβλεφθεί και ότι οι Ρώσοι είχαν σχεδιάσει προσάρτηση της Κρυμαίας. Να ρωτήσω λοιπόν, υπήρχε κάποια πρόβλεψη γι' αυτό. Φαινόταν θα συνέβαινε. Με αναλύσεις που κάνουμε, με όλες τεχνολογίες που έχουμε, δεν ε, είχαμε κάνει κάποια πρόβλεψη ώστε να προστατευτούμε από περαιτέρω παρόμοιες δράσεις που θα επιδεινώσουν την κατάσταση. Κατά πόσο λοιπόν μπορούμε να μιλάμε για τα σενάρια αυτά σε αυτή τη μορφή υβριδικού πολέμου για το μέλλον. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Με την κυρία Χωτέγα επισκεφτήκαμε πρόσφατα την Μολδαβία όπου βλέπουμε ότι υπάρχουν ελπίδες για σταθεροποίηση της πολιτικής κατάστασης στη χώρα. Όμως, δυστυχώς αυτά δεν έγιναν τελικά, παρά τις προσδοκίες και τις ελπίδες. Οπότε, η υπερδυστηνιαρία έγινε κατά κάποιο τρόπο πιο επικίνδυνη από διάφορες απόψεις, γιατί και άλλοι εταίροι μας, όπως οι Ουκρανοί, αντιμετωπίζουν σοβαρά πολιτικά προβλήματα. Οπότε θα ήθελα να μάθω ποιες είναι οι επιπτώσεις όλης αυτής της κατάστασης σε αυτή την ε, περιοχή όσον αφορά το μέλλον, το άμεσο μέλλον. Επίσης να πω ότι ανησυχώ και για άλλες διενέξεις. Εδώ έχουμε ένα σημαντικό ρόλο της γεωργίας και το ρόλο της για την σταθεροποίηση και την ασφάλεια σε κάποιες περιοχές. Εμείς σήμερα δεν εξετάζουμε. Δεν βάζουμε στο μικροσκόπιο τη γεωργία. Θα ήθελα όμως να μάθω πώς αυτή η περιοχή που μας αφορά και μας ενδιαφέρει θα μπορούσε να επηρεαστεί από αλλαγή στην, στην γεωργία. Στον δεύτερο τώρα μιλητή στρέφομαι και να ρωτήσω για το κόστος ή τα κόστη. Μάλλον αριθμοί γενικότερα. 50.000 στρατιώτες έχει η Ρωσία στην περιοχή. Πόσο κοστίζει αυτό για τη συντήρησή τους και μόνο 500 εκατομμύρια. Λέω τώρα έτσι ένα νούμερο. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε αν έχετε κάποια άποψη για το πώς το αντισταθμίζουν αυτό, λόγω ακριβώς της χαμηλής τιμής της ενέργειας αυτή την εποχή. Πώς μπορεί λοιπόν η Ρωσία να επενδύει σε συγκρούσει σε διενέξεις τη στιγμή που οικονομικά τα πράγματα δεν πηγαίνουν και τόσο καλά για αυτούς και πώς αυτά τα κόστη μπορούν να επηρεάσουν την παρουσία της Ρωσίας σε τόσο πολλά επίμαχα σημεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μου δώσατε. Πιστεύω ότι το βασικό ερώτημα είναι τι συμβαίνει σε τελική ανάλυση. Είναι μία μακρά παράδοση τα ρωσικά στρατεύματα στις γειτονικέ χώρες. Είναι φυσιολογικό η ιστορική πραγματικότητα αυτή με την οποία θα πρέπει να συμβιβαστούμε. Το 39 η Ρωσία επέμεινε για τις στρατιωτικές βάσεις στη Φιλανδία και στις Βαλτικές χώρες την επόμενη χρονιά χάρη σε αυτά τα στρατεύματα συνέβησαν τα όσα γνωρίζουμε το 1991 η Ρωσία κατέβαλε κάθε προσπάθεια για να διατηρήσει τα υπάρχοντα στρατεύματα στις γειτονικέ χώρες. Για τις χώρες της Βαλτικής πιστεύω ότι ήταν κομβικό θέμα το να επιτευχθεί η αποχώρηση, αλλά τρία χρόνια αργότερα μετά την ανεξαρτησία του 1994, γιατί αυτό ε, συνδεόταν με τα στρατεύματα από την Ανατολική Γερμανία. Διαφορετικά πολύ φοβάμαι ότι θα είχα να παραμείνει εκεί και εγώ δεν θα ήμουν εδώ σήμερα μαζί σας. Αυτό που με ενδιαφέρει στη δική σας αντίδραση δεν είναι το καινούριο, αλλά το παραδοσιακό μοντέλο Πώς μπορεί, μπορούμε να έχουμε επέκταση της επιρροής κοιτώντας δικαιολογία για την παρουσία στρατευμάτων. Γιατί το ουκρανικό μοντέλο δεν ξέρω αν αυτό που θέλουμε. Το θέμα είναι η πρόκληση κοινωνικών και οικονομικών σειράξεων, το έχουμε θύματα και μετά θα εμφανιστούν κάποιοι άνθρωποι και τα ρωσικά στρατεύματα θα παίξουν το ρόλο ειρηνευτικών δυνάμεων. Πραγματικά στην ουσία προκαλούμε συγκρούσεις και το καλό είναι το να είναι κανείς μέρος της λύσης. Με ενδιαφέρει φέρει ιδιαίτερα η άποψή σας. Χάσαμε το δόγμα το, της Ρωσίας των συμπατριωτών στο εξωτερικό, ήταν στις δεκαετίες του 90. Αυτό ήταν ένα δικαίωμα αυθαίρετο παρέμβαση στις γειτονικέ χώρες προκειμένου να υπερασπιστεί κανείς τους συμπατριώτες του σε μια άλλη χώρα. Και πολύ φοβάμαι ότι η αδράνειά μας, το γεγονός ότι δεν αντιδρούμε σε όλα αυτά, διευκόλυνε τη Ρωσία την έναρξη διάφορων, διάφορων συγκρούσεων και σειράξεων. Ευχαριστώ. Κύριο Στατίνα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Έχω κάποιες ερωτήσεις, αλλά προτού τη θέσω θα ήθελα να καλωσορίσω τους προσκεκλημένους μας και να τους ευχαριστήσω για τις πληροφορίες που μας έδωσαν. Πριν από αυτό, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπε ο κύριος Κάλαν, που ρώτησε, είναι φυσιολογικό αυτό, είναι φυσιολογικό να υπάρχουν ρωσικά στρατεύματα σε ξένες χώρες. Νομίζω ότι εδώ και 100 χρόνια είναι πραγματικά φυσιολογικό. Σκεφτείτε τις, ε, κατοχές που έχουμε ζήσει. Ε, σκεφτείτε το, το Αφγανιστάν, την Απχαζία, τη Φιλανδία. Όλες αυτές οι φάσεις κατοχής από τα ρωσικά στρατεύματα, κατα, κατοχής ε, εδαφών από τα ρωσικά στρατεύματα, φυσικά και μας οδηγούν στο να ε, μιλήσουμε για ρωσικό υπεριαλισμό. Να ρωτήσω κάτι την κυρία Ντίνα. Είπατε ότι ε, υπάρχει πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία. Γνωρίζουμε ότι εκεί δεν υπάρχουν πυρηνικά όπλα, διότι με βάση την σύμβαση της Βουδαπέστης όλα τα πυρηνικά όπλα παραδόθηκαν από την Ουκρανία στην Ρωσία. Ήταν σφάλμα αυτό και αποδεικνύει ότι οι συμφωνίες του 1994 τελικά δεν απέφεραν ε, θετικά αποτελέσματα. Άρα η μοναδική ε, πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα είναι να χρησιμοποιηθούν αυτά από το ρωσικό στρατό. <clears throat> Στην Κρυμαία και στον Ντομπάς πιθανότητα ε, πιθανότατα υπάρχουν, υπάρχουν πυρηνικά όπλα. είμαστε βέβαιοι γι' αυτό όμως. Και ρωτάω διότι εγώ έχω την τσεχοσλοβακική εμπειρία όπου για χρόνια μας ε, έλεγαν ότι ε, ο Ρωσικός στρατός, ο Σοβιετικός στρατός μάλλον, δεν είχε πυρηνικά όπλα στην Τσεχοσλοβασκία. Κάτι που αποδείχθηκε ότι ήταν ψέμα. Άρα στην περιοχή του Ντονμπάς και της Κρυμαίας υπάρχουν, λέτε εσείς, ε, πυρηνικά όπλα αυτή τη στιγμή. Και στο Ναγκόρνο Καραμπάχ έχουν περάσει 25 χρόνια από τότε που διακήρυξε την ε, ανεξαρτησία του. Και 25 χρόνια είναι αρκετά για να αποδείξει μια χώρα ότι πραγματικά αποτελεί μια δημοκρατία πολιτικά, οικονομικά. Άμα πάτε όμως στον αγώνο Καραμπάκ θα, θα διαπιστώσετε ότι η οικονομία είναι πιο ε, ανθυρή από ό,τι της ίδιας της Αρμενίας. Και τρίτον στρατιωτικά. Ε, το Ναγκόρνο Καραμπάκ έχει επιτύχει ήδη δύο στρατιωτικές επιτυχίες. Στις αρχές της του 90, στον πόλεμο του Ναγκόρνο Καραμπάκ και στη συνέχεια σε αυτό που αναφερθήκατε κι εσείς, στον πόλεμο των τεσσάρων ημερών. Και εκεί το Ναγκόρνο Καραμπάχ απέδειξε τη στρατιωτική του ετοιμότητα. Και το ερώτημά μου είναι, δεν είναι πλέον καιρός να αρχίσουμε τη συζήτηση για την αναγνώριση του Ναγκόνο Καραμπάκ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο πρώτα στην, στην κυρία Ντίνερ και στη συνέχεια στον κύριο Μίνουσιαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματα με τη σειρά που μου τέθηκαν. Πρώτο ερώτημα. Γιατί δεν προβλέφθηκαν αυτές οι εξελίξεις. Πρόκειται για ένα από αυτά τα σφάλματα που κάνουν όλοι οι αναλυτές όταν ε, κάνουν μια ανάλυση εκ των υστέρων στην ε, Κρυμαία και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που συνέβησαν εκεί. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία και πάρα πολλοί παράγοντες που δυστυχώς δεν καταφέραμε να τους εντοπίσουμε έγκαιρα. Άμα δείτε τις ε, κοινωνικές εκστρατείες που είχε ε, υλοποιήσει η Ρωσία πριν από μερικά χρόνια ε, υπήρχαν δείγματα. Θα σας πω την εμπειρία μου από το 2012. Τότε υπήρχαν μικρά λεωφοριάκια τα οποία διέσχιζαν ολόκληρη την Κρυμαία και όλα τα λεωφοριάκια αυτά είχαν ε, σημαία με το σταυρό του Αγίου Γεωργίου. Επρόκειτο δηλαδή για, για, για προπαγάνδα. Και κάτι ακόμη, όταν οι Ρώσοι ξεκίνησαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, θα μπορούσαν σε εκείνη τη φάση, βάσει και τις συμφωνίες για το στόλο της Μαύρης Θάλασσας, να χρησιμοποιήσουν, να μεταφέρουν στρατεύματα. Επίσης, χρησιμοποίησαν κενά στην Ουκρανική νομοθεσία με πολύ αποτελεσματικό τρόπο, κάτι που έχει παραδεχθεί και η ίδια η Ουκρανική πλευρά, διότι τα δικά της στρατεύματα δεν, επιτρέπονταν, ε, δεν επιτρεπόταν να χρησιμοποιήσουν όπλα Ακόμη και αν επρόκειτο να δεχθούν επίθεση, αν ε, η επίθεση αυτή γινόταν εκτός στρατιωτικής βάσης. Άρα Υπήρχαν στοιχεία, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να τα εντοπίσουμε. Γιατί απέτυχαν τα think tanks. Ενδεχομένως διότι ε, αναλύσαμε και επικεντρωθήκαμε ε, στις, ε, στις ε, υπαρκτές ε, ένοπλες δυνάμεις και δυστυχώς δεν είχαμε όλα τα στοιχεία στα, στα χέρια μας. Από μια πολωνική σκοπιά, που πολλές φορές επικρίνεται, ε, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ ανησυχητικό το ότι η Ρωσία ενισχύεται. Η μεταρρύθμιση του στρατού που ξεκίνησε το 2009 τώρα έχει αρχίσει να φέρνει αποτελέσματα. Και ο προπολογισμό για τι ένοπλε δυνάμει. Αν έρχεται φέτος για παράδειγμα μόνο σε 5%. Ο Υπουργό Άμυνα προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί στη χώρα μας για να διασώσει τα κονδύλια του προπολογισμού. Επίσης, ε, είναι πολύ σημαντική η στρατιωτική βιομηχανία της Ρωσίας, γιατί θέλει να εξασφαλίσει ότι τα χρήματα που επενδύει θα τις αποφέρουν και κέρδη. Υβριδικός πόλεμος, γι' αυτό μιλάμε, ναι, αλλά υπάρχει και το παραδοσιακό στρατιωτικό, κομμάτι του πολέμου. Χθες δημοσιεύτηκαν ειδήσει για την ε, μεταφορά ε, στρατιωτικού εξοπλισμού από τη Ρωσία στην Ανατολική Ουκρανία. Οι Ρώσοι κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να μας διχάσουν προσπαθούν να μας διχάσουν και εδώ ως Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποκομίσουν ωφέλη. Στην υπερδενιστερία η κατάσταση είναι πάρα πολύ περίπλοκη. Οι αναβληθήσεις προεδρικές εκλογές το απαρχαιωμένο, το παροχημένο σύνταγμα, ε, οι κοινωνικές εντάσεις που υπάρχουν στην ε, υπερδνηστερία περιπλέκουν πολύ τα πράγματα στη συγκεκριμένη περιοχή. Παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψουμε αν η κοινωνία θα κινηθεί προς την κατεύθυνση της Ρωσίας ή προς την κατεύθυνση της Δύσης. Η φτώχεια διευρύνεται και οι Ρώσοι λόγω της κρίσης δεν έχουν τη δυνατότητα να τροφοδοτήσουν την περιοχή αυτή με τον τρόπο που το έκαναν στο παρελθόν. Η Γεωργία. Θα σας πει και ο συνάδελφός μου περισσότερα πράγματα για τη συγκεκριμένη χώρα. τι έτσι αποφασίσαμε να τα χωρίσουμε. Περνώντας σε αυτό που ρωτήσατε για το αν πρόκειται για μια ιστορική πραγματικότητα το να υπάρχουν ρωσικά στρατεύματα σταθμευμένα εκτός Ρωσία. Πράγματι, αυτό είναι ένα ε, φαινόμενο που επαναλαμβάνεται ιστορικά. Όμως το πρόβλημα είναι ότι η ρωσική αυτή παρουσία συμβαδίζει πάντοτε με την, με ισχυρή θέση που θέλει να διατηρεί η ρωσική ε, πλευρά σε μια τέτοια περίπτωση. Γι' αυτό και η Πολωνία πολέμησε μέχρι σε σχάτων ώστε να μην έχει ρωσικά στρατεύματα στο έδαφος της. Προσπαθεί να το αξιοποιήσει αυτό η Ρουσία, βεβαίως. Το χρησιμοποίησαν στην υπερνηστερία, στη σύγκρουση στην, ε, Ουκρανία, στη Λευκορωσία, στον, ε, στον Κάφκασο. Όσον αφορά την προστασία των ε, πολιτών εκτός συνόρων, αυτό είναι εμφανές ότι έγινε στην Απχαζία, στην Νότια Οσετία, όταν ξεκίνησαν τα προβλήματα ε, στη Γεωργία. Γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί ε, τους είχαν αρνηθεί να πάρουν γεωργιανά διαβατήρια και έτσι ήρθε η Ρωσία να τους δώσει διαβατήρια. Και έτσι έχουμε 95% του πληθυσμού στην περιοχή αυτή που ε, κατέχει ρωσικά διαβατήρια. Κάτι που αξιοποίησε η Ρωσία στη διαμάχη και στη διένεξη το ίδιο μπορεί να, πει κανείς ότι αντίστοιχε ε, κινήσεις μπορεί να πει κανείς ότι θα αναλάβει η Ρωσία στην Βαλτική. Η τελευταία ερώτηση αφορούσε τη χρήση των τακτικών όπλων. Από ό,τι γνωρίζουμε από αξιόπιστες πηγές δεν υπάρχουν τακτικά όπλα. Δεν μπορούμε βέβαια να αποκλείσουμε κάτι, ένα τέτοιο ε, ε, δεχόμενο σε ό,τι αφορά τα τακτικά όπλα στη Λευκορωσία γνωρίζουν ότι αρκεί η απειλή. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν βομβαρδιστικά τα οποία έχουν μεταφερθεί στην Κρυμαία, υπάρχουν 122 βομβαρδιστικά Υπάρχουν διάφοροι άλλοι τύποι οπλικών συστημάτων. Οι πύραυλοι είναι συστήματα τα οποία απειλούν όχι μόνο ε, την γύρω περιοχή αλλά και τις βαλτικές χώρες, την Πολωνία, την Τσεχία, τη Σλοβακία. Η Ρωσία δεν χρειάζεται καν να απειλήσει αρκεί να επισύσει την παρουσία αυτών των όπλων ε, και αυτό θα έχει άμεση επίδοση. Ευχαριστώ. Κύριε Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω με τη σειρά που διατυπώθηκαν οι ερωτήσεις. Κυρία Πρόεδρε, έχετε δίκιο όταν λέτε ότι ότι η Ρωσία αποσπά πάρα πολλά ωφέλη από όσα συμβαίνουν στο Κάφκασο. Είναι η αρχαία ή μια παλιά ε, δύναμη η οποία πραγματικά έχει μια προνομιακή σχέση με αυτή την περιοχή. Δύο λόγια για τη Ρωσία και θα αναφερθώ και στο θέμα της στρατιωτικής παρουσίας της. Η Ρωσία στον Κάφκασο βρίσκεται εδώ και τέσσερις αιώνες. Τέσσερις αιώνες επεκτείνεται. 420 χρόνια. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε σε 20 χρόνια μετά τον ψυχρό πόλεμο, 400 χρόνια παρουσίας. Όλοι θα επιθυμούσαμε ως δημοκράτες να δούμε οι χώρες να επιλέγουν οι ίδιες το μέλλον τους. Αλλά βεβαίως υπάρχει η ιστορία και αυτός είναι ο λόγος που η Ρωσία, μεταξύ των άλλων, ακολουθούν μία λογική, λογική ισχύω στην παγκοσμιοποίηση, και αυτό κατάλαβαν οι Ρώσοι, η παγκοσμιοποίηση δεν γνωρίζει ζώνες επιρροής τελείωσε αυτή η λογική του ψυχρού πολέμου. Ενδεχομένω επανερχόμαστε σε μια λογική ψυχρού ε, πολέμου. Αλλά θα πρέπει να συνυπολογίσουμε τη νέα πραγματικότητα. Ε, κυρία Πρόεδρε, οι πηγές που έχουμε σήμερα στην διάθεσή μας μας λένε ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον, κανένα ενδιαφέρον για την Αρμενία σε αυτή την σύγκρουση. Το αντίστατο χρειάζονται status quo, θέλουν να παίξουν το πολιτικό χαρτί και μπορούμε να καταλάβουμε και το Αζερβαϊτζάν. Παράλληλα όμως θα πρέπει να δούμε ποιος κάνει τι. Βεβαίως σύμφωνα με τις πηγές μας, το Ατζερμαϊτζάν είχε 300 νεκρούς, η Αρμενία 100. Η Αρμενία είναι μια μικρή χώρα. Θα πρέπει βεβαίως για να υπάρξει επίθεση, να υπάρξει συγκέντρωση των δυνάμεων. Δεν υπήρχε συγκέντρωση δυνάμεων από πλευράς Αρμενίας και πιστεύω ότι οι διαμεσολαβητές της ομάδας του ΜΙΣΚΑ, τα μέλη της ομάδας του Μίξ να συστήσουν μία επιτροπή έρευνας για να ρηχτεί φως στο τι ακριβώς συνέβη. Δεν υπάρχουν 50.000 στρατιώτες Ρώσοι στο Νότιο Κάφκασο. Δεν υπάρχουν. Πολύ, πολύ, πολύ λιγότεροι. Τα στοιχεία μπορείτε να τα δείτε ε, μπροστά σας τους ε, πληρώνει το Υπουργείο Αμενάσα. Αν δει ε, την πολιτική της Μόσχας και του Πούτιν, καταλαβαίνουμε ότι η προτεραιότητα δίνεται στα ρωσικά, στους στρατιώτες, στα ρωσικά στρατεύματα. Σε ό,τι αφορά το ιστορικό μοντέλο και την ιστορική παράδοση, ε, απάντησα, αλλά με βάση θα επανέλθω και στο τέλος. Σε ό,τι αφορά το θέμα του Ναγκόρκο Νοκαραμπάκ, δεν είμαι εγώ εκείνος που θα αποφασίσω αν θα πρέπει να αναγνωριστεί η ανεξαρτησία του Καραμπάχ. Η διεθνή κοινότητα θα πρέπει να γνωρίζει ποια είναι η καλύτερη εγγύηση για την ειρήνη. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει στον κόσμο μία σύγκρουση όπου οι βασικοί παίκτες, στη συγκεκριμένη περίπτωση οι αρχές του Καραμπάχ, δεν βρίσκονται γύρω από ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων. Δεν μπορεί να υπάρχει ειρήνη στο Καραμπάκ όσο οι αρχές του Καραμπάκ δεν κάθονται γύρω από ένα τραπέζι. Και εδώ επιμένω. Όσο πιο πολλές διεθνείς πιέσεις ασκούνται, όσο πιο πολλές δηλώσεις θα γίνονται για την ειρήνη στο Καραμπάκ τόσο καλύτερο για την επίλυση αυτής της σύγκρουσης. Όσο λιγότερες παρεμβάσεις υπάρχουν, όσο λιγότερη παρουσία πολιτικών υπάρξει στο Γερεβάν, στο ε, Μπακού, τόσο μεγαλύτερος ε, θα είναι ο κίνδυνος πολέμου. Θα πρέπει να υπάρξουν διαδικασίες ρύθμισης προκειμένου να ε, κατευναστεί αυτή η διαδικασία, να, να πνιγεί. Στον πόλεμο των τεσσάρων ημερών πραγματικά με εξέπληξε ο μεγάλος αριθμός παρεμβάσεων, δηλώσεων από τους Ευρωπαίους ηγέτες υπέρ της ειρήνης, ε, υπέρ του τέλους της σύγκρουσης. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το να υπάρχουν αυτές οι δηλώσεις απλά και μόνο γιατί αυτό, με αυτόν τον τρόπο ασκούνται πιέσεις προκειμένου να σταματήσουν αυτή την τρέλα των όπλων και να επιλέξουν τη λογική της ειρήνης. Απέχουμε όμως πολύ ακόμα, απέχουμε πάρα πολύ. Το Καραμπάχ το αναγνωρίζει η Καλιφόρνια, οι ορισμένα ομόσπονδα κράτη. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ε, ορισμένοι θεωρούν ότι μπορεί να υπάρξει αναγνώριση και στην Γαλλία και στην Ευρώπη. Υπάρχουν περιοχές, υπάρχουν χώρες που θέτουν το ερώτημα. Συνεπώς θα πρέπει να τα δούμε τα πράγματα με έναν διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, ποιον ωφελεί αυτή η σύγκρουση τους εθνικιστές και από τις δύο πλευρές, ε, τους, εθνι, ε, εθνικές του, του Μπορ και τη Ρωσία βέβαια. Και ευνοεί τη Ρωσία. Πιστεύω ότι είτε μιλάμε για την Ουκρανία, είτε για την Μολδαβία, είτε για τον Νότιο Κάυκασο όλοι έχουν άδικο στην περίπτωση αυτή. Οι Ουκρανοί έχουν άδικο γιατί εδώ και 25 χρόνια κάνουν ένα και μοναδικό πράγμα. Κατέστησαν τη χώρα τους μία γεωπολιτική αξία. Δίχως να θέσουν το ερώτημα ότι θα έπρεπε να έχουν ένα κράτος. Έδωσαν γεωπολιτικό χαρακτήρα στη χώρα τους. Οι Ρώσοι έχουν άδικο. Έχουν άδειο γιατί δεν ξέρουν να κάνουν τίποτα άλλο από το να παίζουν, να ασκούν εξουσία. Αυτό είναι δράμα. Και εμείς οι δυτικοί έχουμε άδικο. Δηλαδή θέλουμε να επεκτείνουμε τις αξίες μας σε όλο τον κόσμο. Ωραία. Όταν όμως υιοθετούν τις αξίες μας χώρες όπως η Υγεία, η Ουκρανία και οι χώρες αυτές εξ ονόματος αυτών των αξιών ε, αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη Ρωσία, εμείς τους γυρίζουμε τις πλάτες και τους λέμε βγάλτε τα πέρα μόνοι σας. Ε, είναι πραγματικά εγκληματικό αυτό. Αυτό θα το γράψει η ιστορία, γιατί εμείς οι Δυτικοί μπορούμε να εγγυηθούμε την ειρήνη σε αυτές τις χώρες. Δεν μπορούμε όμως να εγγυηθούμε την ασφάλεια. Δεν θα υπάρξει ένας ευρωπαϊκός στρατός έτοιμος να πάει στην Κρυμαία ή στον Κάφκασο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποια ευθύνη και η ευθύνη αυτή είναι συλλογική. Ενδεχομένω θα πρέπει να επανεξετάσουμε το διεθνές σύστημα. Και βεβαίως αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Τώρα, θα ήθελα να τελειώσω αναφερόμενος στο βασικό θέμα που έχει σχέση με την περιοχή του Καυκάσου. Εδώ ο βασικός εχθρός, και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα μοντέλο soft power Διακρατική. Ο κίνδυνος είναι ο εθνικισμό αυτέ αυτές τις χώρες και κατ' επέκταση ε, η ε, απουσία ενσυναίσθησης για τον άλλον. Βλέπουν τον άλλον ως κατώτερο. Και αυτό είναι το βασικό διακύβευμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Ευχαριστώ. Unfortunately... Ευχαριστώ. Έχει περάσει ο χρόνος μας. Στέτιανα και Βότσον, παρακαλώ σύντομη να είστε στις ε, ομιλίες Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για αυτή την εξαίρεση. Να πω ότι με τον προλήσαντα συμφωνώ απολύτως με αυτά που είπε. Ότι πράγματι θα πρέπει να παρανεύουμε στις πολιτικές για τον Αγκόρνο Καραπάχ. Εγώ επισκέφθηκα αυτή την περιοχή μετά το σύντομο πόλεμο. Πήγα στο κοινοβούλιο των αγώνο Καναπάχ και συζητήσαμε τη δυνατότητα βουλευτέ του να έρθουν να επισκεφτούν εδώ το Ευρωκοινοβούλιο. Να του ακούσουμε, να δούμε τι έχουν να μα πούν και είναι έτοιμοι να το πράξουν. Υποβάλλω λοιπόν την ιδέα αυτή να γίνει αυτή η επίσκεψη και να διερευνήσουμε κατά πόσο μπορεί να γίνει σύντομα. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Υποσχέθηκα να σας το λόγο. Δυστυχώ ο χρόνος μας όμως έχει τελειώσει. Κλείνουμε λοιπόν με αυτό το σημείο της ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ του εισηγητέ μας για τις πολύ ενδιαφέρουσε εισηγήσει του. Και βεβαίω θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για αυτό το θέμα στο μέλλον. Ευχαριστώ. I kindly ask... Uh, Σας ζητώ, αγαπητά μέλη και υπόλοιποι συμμετέχοντες, να καθίσετε.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 καθίσετε γρήγορα όλοι οι παρόντες εδώ στην αίθουσα Okay. Next. Ωραία. Επόμενο σημείο της σημερινής διάταξη. Σύντομο σημείο, στην επόμενη, αρκετά τεχνικό βέβαια, είναι η ενημέρωση για την αποστολή μας στην Γεωργία. Ο κύριος σκοπός της αποστολής μας ήταν η αποτίμηση των δράσεων της αποστολής που πήγε στη Γεωργία της EUMM αποστολής εποπτείας επισκεφθήκαμε δύο υπηρεσίες ΣΕΤΑ και ΓΚΟΡΙ σε αυτές τις τοποθεσίες και έχουμε θαυμάσει αρκετά βέβαια τεχνικές επισκοπήσεις και τις επισκέψεις και στο Τζιακάουσκας ε, είναι αυτός που θα μας κάνει την παρουσίαση τη δεύτερη φορά μάλιστα μπορέσαμε να συναντήσουμε τον επικεφαλής της αποστολής Είχαμε το κριτήριο για Σκάουσκας που μας ενημέρωσε για τις δράσεις της UMM. Εγώ είχα επισκεφτεί βέβαια την υπηρεσία αυτή νωρίτερα στην αρχή του έτους αλλά βλέπουμε ότι τώρα αυτή η επίσκεψη μας επέτρεψε να έχουμε μια ευρύτερη εικόνα για τις δράσεις της αποστολής αυτής. είχαμε και ημερήσιες περιπολίες κατά τη διάρκεια αυτής της αποστολής των παρατηρητών όπου επισκεφθήκαμε και το διοικητικό, να το πω έτσι, σύνορο στην Νότια Σετία και στην Τυφλίδα ώστε να δούμε ακριβώ πώς εξελίσσεται η διαδικασία χαράξη των συνόρων. Βλέπουμε να υπάρχουν χωριά τα οποία έχουν χωριστεί στη μέση. Βλέπουμε να υπάρχουν μέρη όπου οι ρωσικές δυνάμεις κάνουν τις ε, ασκήσεις στην επικράτηση της Οσετίας δηλαδή. Είχαμε επίσης και πολύ ενδιαφέρουσες διμερείς συναντήσεις υψηλού επίπεδου με τον πρόεδρο της Γεωργίας, τον πρωθυπουργό της Γεωργίας, υπουργούς της Γεωργίας, συγκεκριμένα υπουργός άμυνας, Υφυπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό για την ε, ενσωμάτωση, όπως επίσης και με κιό συναντήσαμε. Εγώ και ο Μάρκολ Γκάλερ μπορέσαμε επίσης να επισκεφτούμε υψηλόβαθμους πολιτικούς που κρατούνται στη φυλακή στην Γεωργία. Η Βαλαμάρ φίλοι την πρώην Πρωθυπουργό, πρώην Υπουργό Αμινάσα Αχαλάγια και τον πρώην Δήμαρχο Ουκλάβα της Τυφλίδας. Ποια είναι η κατάσταση τώρα στη Γεωργία. Ιδιαίτερα όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα. Να πούμε καταρχάς ότι οι δράσεις της EUMM, της αποστολής παρατηρητών, ήταν πολύ θετικές. Συζητήσαμε την ανάγκη βέβαια για αλλαγές σε τομείς όπως η δικαιοσύνη. Καταγράψαμε βέβαια και τις προσπάθειες που γίνονται στα πλαίσια της μεταρρύθμισης στο δικαστικό τομέα. Και συζητήσαμε καταστάσεις όπως αυτές που αφορούν την φυλάκιση βέβαια μελών της αντιπολίτευσης. Είπαμε και σε συζητήσεις με τις ΜΚΟ ότι θα πρέπει να υπάρχει πλουραλισμός στα ΜΜΕ της Γεωργίας και κατά το τέλος της αποστολής είχαμε μια ενημέρωση από τον Υπουργό Εσωτερικών και μπορούσαμε να μεταφέρουμε στα μέσα την ε, συνένεση των εκπροσώπων των τεσσάρων μεγαλύτερων πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συμμετείχαν στην αποστολή αυτή επειδή βέβαια εμεί εκπροσωπούμε τέσσερις μεγάλες πολιτικές ομάδες και ομονοήσαμε συμφωνήσαμε απόλυτα στο να υπάρχει άνοιγμα του καθεστώτος της Γεωργίας το ταχύτερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από τις εκλογές. Ελπίζουμε λοιπόν να υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα και στη συζήτηση στο Συμβούλιο σε σχέση με αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις για αυτό το ζήτημα, γιατί εγώ με αυτά που σας είπα μόλις τώρα τέλειωσα, δεν ξέρω αν έχετε εσείς παρατηρήσεις. Ο κ. Τρογεύσκη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ένα ερώτημα προς εσάς, κυρία Πρόεδρε, γιατί ξέρω ότι συναντηθήκατε με κρατούμενους Ποιος ήταν ο χαρακτήρας αυτών των ε, συναντήσεων. Ε, το κομμάτι αυτό δεν ήταν επίσημο τμήμα της αποστολής, γιατί οι εξουσιοδοτήσεις δίνονται ατομικά. Οπότε εγώ ατομικά ζήτησα εξουσιοδότηση να δω αυτούς τους κρατόμενους. Πήγαμε εγώ και ο κύριος Γκάλε και δεν ήταν η πρώτη φορά. Είχαμε ε, ξαναεπισκεφτεί πολιτικούς κρατούμενους ε, στις φυλακές της χώρας στο παρελθόν. Αν θέλετε να ακούσετε την εντύπωση που αποκόμισα, θα χρειαστούμε πάρα πολύ χρόνο. Ε, η ε, χθεσινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όσον αφορά τον κύριο Μεραβισβίλη, πρώην Πρωθυπουργό της Γεωργίας, αποδεικνύει ότι κάποιες από τις διαδικασίες που εφαρμόστηκαν στην περίπτωσή του είχαν σαφή πολιτικό χαρακτήρα. Και αυτό αναφέρεται ρητός στην απόφαση του δικαστηρίου. Ότι πολλές από τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ε, έγιναν κατά παράβαση του νόμου. Και αυτό σημαίνει ότι διώχθηκε ο άνθρωπος αυτός λόγω του ότι ήταν επικεφαλής της αντιπολίτευσης και επειδή ήταν υποψήφιος για θέση στο κοινοβούλιο. Σκοπός του ήταν να μεταρρυθμιστεί η εκλογική διαδικασία. Και όλα αυτά τα αναφέρει στην, ε, στην απόφασή του και στο σκεπτικό της απόφασης που συναδεύει την απόφαση αυτή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σε κάθε περίπτωση, για μένα ήταν μια προσωπική, αν θέλετε, ε, επιλογή, κίνηση και το κάνω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί γνωρίζει όλος ο κόσμος τον σεβασμό που τρέφω για τη Γεωργία και για τον γεωργιανό λαό, ανεξαρτήτως του ποιος είναι στην κυβέρνηση. Πιστεύω ότι η Γεωργία ανήκει στο δυτικό κόσμο και θα πρέπει αυτό να γίνει το συντομότερο δυνατό, καθώς πρόκειται για μία από τις χώρες με τις οποίες έχουμε την ισχυρότερη συνεργασία, ιδιαίτερα σε ζητήματα ασφαλείας στο πλαίσιο της αποστολής μας, ε, ε, την, ίδια, την ίδια περίοδο μάλλον ε, που έγινε η αποστολή μας, έγιναν και στρατιωτικές επιχειρήσεις Αμερικανών, Βρετανών και Γεωργιανών. Και εμείς είχαμε με αφορμή αυτή την στρατιωτική άσκηση τη δυνατότητα να συζητήσουμε και με νατοικούς αξιωματούχους στην Γεωργία. Ξέρουμε ότι η Γεωργία ε, έχει και άλλες μορφές συνεργασίας και γνωρίζουμε ότι παρά την τωρινή της ε, κυβέρνηση ε, πρόκειται για μια χώρα η οποία είναι αποφασισμένη να ακολουθήσει στο δρόμο της ανάπτυξης. Μετά την συνάντησή μας με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας μας παραδόθηκε από τον ίδιο μάλλον μία ε, πολύ ολοκληρωμένη έκθεση όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και τις αντίστοιχες προσπάθειες που καταβάλλονται στη χώρα και τον ε, σχετικό οδικό χάρτη, ο οποίος και θα επιτρέψει στη χώρα να ε, αποκτήσει ένα νέο καθεστώς απελευθέρωσης των θεωρήσεων. Ο κύριος Στατίνα. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να σας πω ένα πράγμα. Χθες στην Επιτροπή ΑΦΕΤ συζητήσαμε το θέμα της ε, απελευθέρωσης των θεωρήσεων για την γεωργία. Οι περισσότεροι από αυτούς που πήραν το λόγο χθες ήταν υπέρ της επιτάχυνσης και όχι της επιβράδυνσης των διαδικασιών. Αυτή ήταν η άποψη της Επιτροπής ΑΦΕΤ, η οποία ταυτίζεται με την άποψη της κυρίας Πρόεδρου. Η Γεωργία είναι μέρος της Ευρώπης και νομίζω ότι μία κίνηση προς την κατεύθυνση των θεωρήσεων θα ήταν κάτι πάρα πολύ θετικό. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να κλείσουμε το σημείο αυτό της ημερησίας διάταξης. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να συγχωρήσετε την αναχώρησή μου. Έχω κάποιες άλλες σημαντικές συνεδράσεις και θα παρακαλούσα τον κύριο Στατίνα να αναλάβει την Προεδρία. Αύριο έχουμε να συζητήσουμε δύο σημαντικά σημεία στην μερισία διάταξη συμπεριλαμβανομένων και συναντήσεων ε, με προσώπους του ΝΑΤΟ και έλασον και όχι ελάχιστον την παρουσίαση του κυρίου Σολάνας και θα είναι βεβαίως και ο ίδιος παρόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, την ετοιμή για μένα η ανάληψη της Προεδρίας αυτής της συνεδρίασης. Να περιμένουμε ένα-δυο λεπτά για τους καλεσμένους μας για να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Σε λίγα λεπτά ξεκινήσουμε. Eh, λοιπόν, ας περάσουμε λοιπόν στο τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης για σήμερα. Εξίσου ενδιαφέρον και με τα θέματα που συζητήσαμε πριν, αλλά και το πρωί. Και μιλούμε για τις υβριδικές απειλές. Υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια βεβαίως τα είχαμε, υπήρχαν ακόμη και στους ε, πολέμους του Μεσαίωνα. Αλλά το τελευταίο διάστημα ο όρος αυτός ακούγεται όλο και περισσότερο σε σχέση με την Ουκρανία. Δεν αφορά όμως μόνο την Ουκρανία, αλλά αφορά συνολικά και την, ε, και την καταπολέμηση, τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. Πρόκειται για μια απειλή που για την αντιμετώπιση της αποτελ, απαιτούνται, απαιτείται ενότητα των, ε, εδώ, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και αξιοποίηση όλων των, εσωτερ, των ε, εργαλείων εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής που έχουμε στη διάθεσή μας. Τον Μάρτιο του 2016 είχαμε ήδη συζητήσει το θέμα των υβριδικών πολεμικών απειλών. Επίσης, εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση για, τον, για το είδος των υβριδικών πολέμων και με τις δυνατότητες αντιμετώπισης των υβριδικών αυτών απειλών. Οι εξελίξεις είναι σχετικά πρόσφατες. Ωστόσο, έχουν περάσει κάποιοι μήνες από τότε που εκδόθηκε αυτή η κοινή ανακοίνωση και θα θέλαμε να δούμε ποια ήταν η απήχηση της. Γι' αυτό και θα μιλήσουμε με τον κύριο Πιέρ Ντελσό, αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης GROW της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον κύριο Γκάμπορ Ικλόντι, Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κρίσεων και Προγραμματισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και καλωσορίζω και τον κύριο Χούζε, τον αναπληρωτή ε, διευθυντή ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Ποιος θα ήθελε να ξεκινήσει. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Λοιπόν, μια και είμαι εγώ ο πρώτος που κατέφτασα, ξεκινώ εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας να συζητήσουμε εδώ αυτή τη σημαντική ανακοίνωση της Επιτροπής και της ΕΕΔ για τις ευρυδικές απειλές. Σήμερα ε, μάθαμε ότι υπάρχουν νέες απειλές επιθέσεων τρομοκρατικού χαρακτήρα στην Γαλλία και στο Βέλγιο και για τα κράτη-μέλη, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βεβαίω για του πολίτε, το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και να, πάμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση ασφάλεια στην Ευρώπη. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλέ διαστάσει και πάρα πολλέ πτυχέ που πρέπει κανεί να εξετάσει. Είναι σαφέ ότι από τη σκοπιά τη επίτροπή το ζήτημα αυτό είναι θεμελιώδου σημασία, και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνά από τα χέρια μα προκειμένου να εξεύρουμε μια λύση. Ενημερωτικά και προτού περάσω στην ανακοίνωση για τις ευρυδικές απειλές να σας πω ότι η Επιτροπή πρόκειται να εκδώσει και ανακοίνωση για ένα σχέδιο δράσης για την άμυνα γιατί θεωρούμε ότι και η άμυνα είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό και η ανακοίνωση αυτή θα εκδοθεί, το σχέδιο δράσης μάλλον θα υιοθετηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Για τις υβριδικές απειλές. Βλέπετε εμείς οι τρεις ομιλητές ε, το αποδεικνύουμε με την παρουσία μας εδώ, ότι πρόκειται για μια κοινή άσκηση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ε, άμυνας. Σε όλα τα στάδια συνεργαζόμαστε, γιατί υπάρχει ένα σημαντικό μήνυμα το οποίο πρέπει να αποστείλουμε και αυτό είναι ότι απαιτείται συνεργασία. Τα τρία θεσμικά όργανα λοιπόν που βρίσκονται εδώ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη. Χωρίς ενότητα δεν θα τα καταφέρουμε. Χρειάζεται να βρούμε έναν τρόπο συνεργασίας. Αν δείτε την ίδια την ανακοίνωση και αυτό που έχουμε εγκρίνει, ε, θα ήθελα να σας ε, να ε, παρουσιάσω κάποια στοιχεία σημαντικά. Έχουμε προσδιορίσει τέσσερις τομείς δράσης. Πρώτον, χρειάζεται να καταλάβουμε να κατακτήσουμε μια κοινή αντίληψη για τις υβριδικές απειλές. Αυτό είναι θεμελιώδους σημασίας αν θέλουμε να εντοπίζουμε απειλές υβριδικού χαρακτήρα. Θα, θα δώσω το λόγο στον Γκάμπορ και ο Γκάμπορ θα σας εξηγήσει αργότερα τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Δεύτερη ε, θεματική ενότητα. Πρέπει να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητά μας. Θα επανέλθω σε αυτό. Τρίτο στοιχείο. Πρέπει να οργανώσουμε την απάντησή μας στις ευρυδικές απειλές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση ε, άμεσων απειλών. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε στα χέρια μας τα κατάλληλα μέσα για να ανταποκριθούμε σε περίπτωση ε, κρίσεων. Και τέλος, προτείνουμε να δημιουργηθεί ε, μια ειδική μορφή συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ για τις τρομοκρατικές απειλές. Στη δική μου ομιλία θα επικεντρωθώ στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας που είναι θεμελιώδους σημασίας διότι γνωρίζετε ότι οι, ε, οι ευρετικές απειλές ε, έχουν ως στόχο να εντοπίσουν τα ευάλωτα σημεία μας. Θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα συγκεκριμένων στρατηγικού χαρακτήρα τομέων. Τι πρέπει να κάνουμε. Να δούμε την κυβερνοασφάλεια. Πρέπει να δούμε την ε, κρίσιμη ε, υποδομή στην ενέργεια στην, και στις μεταφορές. Πρέπει να πάρουμε συγκεκριμένα μέτρα για να ε, προστατεύσουμε τα χρηματοπιστωτικά συστήματα και να ε, μπορέσουμε να αποκτήσουμε μέσα για την απόκρουση της ριζοσπαστικοποίησης. Πρέπει επίσης να ε, βρούμε, να εντοπίσουμε τους πόρους χρηματοδότησης των υβριδικών απειλών. Να πω όμω ότι δεν είναι όλα τα πράγματα καινούργια. Ούτε ξεκινάμε από το μηδέν. Έχουμε μια σειρά από ευρωπαϊκέ πολιτικέ που έχουν ω στόχο την ενίσχυση τη ανθεκτικότητας, τη πρόληψη και τη ασφάλεια. Δεν θα σα τι παρουσιάσω, αλλά υπάρχει πραγματικά ένα πολύ μεγάλο αριθμό μέτρων και πολιτικών. Ένα πράγμα όμω είναι πολύ σημαντικό που πρέπει να το τονίσουμε. Οι βρεδικέ απειλέ έχουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα και ένα από τα στοιχεία που χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε άμεσα είναι να σταματήσουμε την σιωπή. Πρέπει να ε, δράσουμε με συνέργειες και διατομιακά να αποκτήσουμε μια ολιστική προσέγγιση προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις υβριδικές απειλές όταν αυτές εμφανίζονται. Ένα πρώτο στοιχείο που αντιμετωπίζουμε, ε, που θεωρούμε ότι είναι σημαντικό. Δεύτερον, πρέπει να προσδιορίσουμε επιπρόσθετες προτάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της ανθεκτικότητάς μας, ιδίως όσον αφορά τις υποδομές μας. Και τρίτη διάσταση είναι ότι χρειάζεται να ενισχύσουμε την δυνατότητά μας, την ικανότητά μας να ανταποκριθούμε σε περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος δεχθεί επίθεση και θα, πρέπει να μπορούμε να χρησιμοποιούμε και να αξιοποιούμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στην ε, διάθεσή μας και όλα όσα προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας. Κυρίες και κύριοι, η ανακοίνωση βεβαίως ε, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα και όπως είπα αποτελεί έργο συνεργασίας των τριών θεσμικών οργάνων. Αλλά δεν είναι το τέλος του δρόμου. Αντιθέτως, βρισκόμαστε στην αφετηρία και το βασικό στοιχείο είναι πώς θα υλοποιήσουμε τις 22 δράσεις που περιγράφονται στην ανακοίνωση αυτή. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλοι μας από τη σκοπιά του ο καθένας θα ε, εργαστεί στο μέτρο των δυνατοτήτων του προκειμένου να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί από κοινού αυτές τις υβριδικές απειλές οι οποίες δεν θα μας περιμένουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα σε όλους σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, ευκαιρία που μου δώσατε να σας συναντήσω και να μιλήσουμε για τα τόσο σημαντικά αυτά θέματα. Θα ήθελα να τονίσω ότι βρισκόμαστε στην αρχή και όχι στο τέλος του δρόμου. Η εφαρμογή είναι κάτι που μένει ακόμα να γίνει. Μιλήσαμε, μιλάμε πολύ για τις υβριδικές απειλές. Έγινε μία λέξη του σειρμού, θα έλεγα χρησιμοποιείται από ακαδημαϊκούς, από εφημερίδες ευραίως. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο υβριδικές ε, απειλές. Γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να κολλάμε ταμπέλες και να λέμε ότι πρόκειται περί υβριδικής απειλής. απειλές ε, ή προβλήματα παροχής ενέργειας δεν είναι κατά ανάγκη υβριδικές απειλές. Είναι ο συνδυασμός διαφορετικών διάφορων συγκαλυμμένων και μη συγκαλυμμένων καταστάσεων συμβατικών και μη συμβατικών, καταναγκασμός και μη καταναγκασμός, πολιτικός και στρατιωτικός. Είναι δηλαδή ένα συνδυασμός διαφόρων στοιχείων. Αν ισχύσει με ένα κεντρικά σχεδιασμένο τρόπο προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι, αυτό αποσταθεροποιεί τα θύματα των επιθέσεων. Και στην περίπτωση αυτή θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για υβριδικές απειλές. Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό των υβριδικών απειλών είναι ότι αλλάζουν, προσαρμόζονται και εξαρτάται από τις ε, απαντήσεις που δίνουμε κάθε φορά. Αυτές οι υβριδικές απειλές προήλθαν από πολλές μεριές το παρελθόν το κοινό ανακοινωθέν προσπαθεί να επιληφθεί και των δύο απειλών, μόνο ότι η φύση τους είναι διαφορετική, αλλά ε, υπάρχουν ορισμένα κοινά στοιχεία. Έχουμε τις ε, απειλές, ας πούμε, που προέρχονται ε, εξανατολών. Ένα ε, χαρακτηριστικό αυτών των απειλών είναι ότι έχουν στη βάση τους ε, το γεγονός ότι είμαστε ευάλωτοι. Ενδεχομένως μπορεί να αφορά τον ευάλωτο χαρακτήρα των κοινωνιών ή τον ευάλωτο χαρακτήρα των υποδομών μας ή των θεσμών μας, των θεσμικών μας οργάνων και στόχος είναι αυτός ο ευάλωτος χαρακτήρας. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό των υπηρετικών απειλών είναι ότι προσπαθούν πάντοτε να δημιουργήσουν ένα αμφίσιμο περιβάλλον, να μην ξέρει κανείς τι συμβαίνει, τι είναι αυτά τα πράσινα ανθρωπάκια. Η δημιουργία λοιπόν της αίσθησης ευαλωτότητας διευκολύνει κάποιον να, διακράψει, να διαβράξει ένα δίκημα και καθιστά πιο δύσκολη τη λήψη αποφάσεων. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι οι υβριδικές απειλές προσπαθούν να κρατηθούν κάτω από ένα κατόφλι, να μην φτάσουν σε ένα όριο που θα προκαλέσει μια αντίδραση κάθε φορά βεβαιώνονται ότι παραμένουν κάτω από τον ουδό, κάτω από ένα ε, κατόφλι. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι πολύ συχνά οι υβριδικές απειλές προέρχονται από καμπάνιες παραπληροφόρησης. Δηλαδή, δημιουργείται μία εικονική πραγματικότητα η οποία προσπαθεί να σας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Εδώ δεν μιλάμε για ένα πραγματικό κόσμο, μιλάμε για μια εικονική πραγματικότητα. Τι θα μπορούσαμε λοιπόν να κάνουμε. Το πρώτο είναι να γνωρίζουμε σε ποια σημεία βρισκόμαστε ευάλωτοι. Εύκολα να το λες, δύσκολο να το κάνεις, γιατί ακόμα και στις ίδιες χώρες, τις ίδιες χώρες είναι δύσκολο να γνωρίζουμε σε ποια σημεία βρισκό, είμαστε ευάλωτοι. Αλλά αν θέλουμε πραγματικά να βρούμε αλληλεγγύη σε μια ευρύτερη κοινότητα, θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σχετικά με το ποια είναι τα σημεία που είμαστε ευάλωτοι. Μέσω της εφαρμογής ε, ε κοινών ανακοινοθέντων, θα προσπαθήσουμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Θα γίνουν έρευνες σχετικά με τον εντοπισμό αυτών των σημείων που είμαστε ευάλωτοι. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα του τι συμβαίνει και το τι επέρχεται. Αυτό επίσης έχει σχέση με την συνδυτότητα. Πολύ συχνά μπορείτε να εντοπίσετε μερικούς δείκτες που μας λένε ότι υπάρχει μια τρέχουσα υβριδική δραστηριότητα και υπάρχουν σημάδια που προέρχονται από διάφορες περιοχές. Τότε μπορεί κανείς να αρχίσει να υποψιάζεται ότι υπάρχει κάποιος εγκέφαλος από πίσω και ότι κατευθύνονται κεντρικά όλες αυτές οι δραστηριότητες. Το πιο σημαντικό για να αντισταθμιστούν αυτές οι δράσεις είναι το να αυξήσουμε την ανθεκτικότητά μας. Και μιλάμε για την κοινωνία, για τις υποδομές, για τους διάφορους φορείς. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά η Επιτροπή θα μπορούσε να δώσει ιδιαίτερη στήριξη στα κράτη-βέλη προκειμένου να γίνει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της πρόληψης και της αποτροπής αυτός ο όρος δεν χρησιμοποιείται ε, εκτενώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εμείς έχουμε αρκετούς ε, αποτρεπτικούς μηχανισμούς στην παρέτρα μας. Έχουμε εργαλεία, έχουμε μέσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να αποθαρρύνουμε κάποιον ε, από τον δράστη, από τον δυνητικό δράστη. Βεβαίως, αν αποτύχει η παρέμβαση, το επόμενο βήμα είναι η αντίδραση, η απάντηση. Και εδώ η κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να επιδείξει αλληλεγγύη. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει διαδικασία λήψης αποφάσεων. Είναι ένα αμφίσιμο περιβάλλον, δεν ξέρει κανείς τι συμβαίνει. Παρόλα αυτά, οι λαμβάνοντες αποφάσεις θα πρέπει να δράσουν άμεσα και με αποφασιστικότητα. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τους λαμβάνοντες αποφάσεις να καταλάβουν έτσι ώστε να μπορέσουν άμεσα να πάρουν αποφάσεις. Δεν αντιμετωπίζουμε τις ε, υβριδικές απειλές απομονωμένοι. Δεν είμαστε ρομπινσόνες κρούση. Συνεπώς, ενδεχομένως θα το έχετε δει στο κοινό ανακοινωθέν, ότι δίνεται μεγάλη σημασία στη συνεργασία μεταξύ Ατλαντικής Συμμαχίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δύο οργανισμοί θα πρέπει να προσπαθήσουν από κοινού να αναπτύξουν μηχανισμούς και να συνεργαστούν και σε επίπεδο αντίδρασης, αποτροπής και συνειδητότητας. Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων το Μάιο του 2015 συζήτησε αυτά τα θέματα και μας ζητήθηκε να αναπτύξουμε μέτρα προκειμένου να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν τις υβριδικές απειλές ε, όχι μόνο τις χώρες μέλη αλλά και τις χώρες εταίρου και βεβαίως να αυξηθεί η ανθεκτικότητά τους. Νομίζω ότι υπάρχει μια ανάγκη διάκριση των κρατών μελών και των ε, εταίρων. Θα πρέπει να συνεργαστούμε πάρα πολύ στενά, αλλά βρισκόμαστε μόνο στην ε, αρχή της πορείας μας. Όλα αυτά ε, κοινοποιήθηκαν στα κράτη-μέλη. Η εφαρμογή θα γίνει μέσω της, ε, των Επιτροπών Μονίμων Αντιπροσώπων ή θα συντονιστούν από τα κορεπέρα. Είναι πολύ σημαντικό δούμε το θέμα από πολλές οπτικές γωνίες, γιατί η ασφάλεια είναι καθοριστικός παράγοντας σε αυτό που θα κάνουμε εδώ. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ρόλο ε, της ΙΕΣ ε, θα δημιουργηθεί ένα συγκεκριμένο ένα κύτταρο θα δημιουργηθεί στο κέντρο πληροφοριών, στο ΙΕΣ, θα συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη, με μερικές από τις χώρες εταίρου, θα συγκεντρώνει πληροφορίες, θα τις ταξινομεί τις πληροφορίες, αναλύει αυτές τις πληροφορίες. Και θα προσπαθεί να εντοπίσει εάν είμαστε εκτεθειμένοι σε μία απειλή, σε μία ευρυδική δράση και μετά θα μπορεί να κάνει συστάσεις σε ό,τι αφορά μία πορεία ή μία δράση που θα μπορούσε να αναλυθεί προκειμένου να σταματήσει μία ενέργεια ή να αμβληθούν οι επιπτώσεις της. Θα δημιουργηθεί ένα κέντρο και σκοπό θα έχει διεξαγωγή ερευνών ή κατάρτιση η άσκηση στον τομέα των υβριδικών ενεργειών, των υβριδικών απειλών. Ήδη αναφέρθηκα στο θέμα της συνεργασίας ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δύο οργανώσεις θα συνεργαστούν έτσι ώστε να υπάρχει μία κοινή εικόνα, ένα κοινό σημείο κίνησης. Δεύτερον, θα πρέπει να εναρμονίσουμε τους μηχανισμούς αντίδρασης για να έχουμε τη βεβαιότητα ότι μπορούμε να δράσουμε άμεσα παρέχοντας τη βέλτιστη των υπηρεσιών στα κράτη-μέλη. Ο κυβερνοχώρος είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις δύο οργανώσεις να συνεργαστούν και τέλος στρατηγικές και επικοινωνία προς το κοινό μας, προς τον αντίπαλο. για να πούμε τι ακριβώς ε, συμβαίνει με σαφήνεια και για να πούμε ότι είναι σημαντικό να παραμείνουμε ενωμένοι. Ε, Επιτρέψα μου να αναφέρω τρεις ε, τομείς που μας προβληματίζουν. Το πρώτο, όπως είπαμε, είναι ο ευάλωτος χαρακτήρας αυτού του θέματος είναι σημαντικό να αποκαλύψουμε μάλλον τα ευάλωτα σημεία μας. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι για ένα κράτος να το κάνει. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τα ευάλωτα σημεία μας. Υπάρχουν χώρες που εκτίθενται άμεσα σε αυτές τις υβριδικές απειλές. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει διαφάνεια. Ανταλλαγή πληροφοριών ως είναι ένας άλλος δασικός τομέας. Ε, επειδή πολλές ε, πληροφορίες είναι ε, εμπιστευτικές, μερικές φορές είναι θέμα κουλτούρας. Να υπάρξει δηλαδή μια κουλτούρα σε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ότι μπορούμε να δουλεύουμε έχοντας τη βάση, έχοντας τα χέρια μας εμπιστευτικές πληροφορίες. Αν υπάρξει κάποια διαρροή, βεβαίω αυτό είναι πρόβλημα. Θα πρέπει να αλλάξουμε την κουλτούρα μας, όπως είπαμε μέσα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αλλά και μέσα στα ίδια τα κράτη-μέλη. Αυτό λοιπόν που χρειαζόμαστε είναι μια κυβερνητική προσέγγιση. Όχι μόνο θέματα ενέργειας ε, ή άλλα θέματα. Θα πρέπει αυτά να τα δούμε σε όλη την Ευρώπη. Αυτή είναι η ίδια η φύση των ε, ιδρυτικών απειλών. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω το θέμα της αλληλεγγύης, που είναι ένα βασικό στοιχείο. Αν διαβάσετε το κοινό ανακοινωθέν θα διαπιστώσετε ότι προτείνεται κάποια δάση στην, σε ό,τι αφορά το άρθρο 42,7 και το άρθρο 222 των συνθήκων. Πώς λοιπόν η αλληλεγγύη μέσα στην ευρωπαϊκή κοινότητα θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε περίπτωση που βρεθούμε αντιμέτωποι με μία υβριδική επίθεση ή σε περίπτωση που υπάρχει υβριδική απειλή. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα, τελευταίος, ο κύριος Γκος από την Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων και Πραγματισμού Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρόλο που είμαστε μέρο αυτής της διαδικασία της πολιτικής, σας ευχαριστώ που μας καλέσατε για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Το κοινό πλαίσιο αποτελεί το καλύτερο μέσο για να αντιμετωπίσουμε τις απειλές και να επιφέρουμε αυτή την αθεκτικότητα που λέγαμε. Εγώ θα επικεντρωθώ στα αποτελέσματα του κοινού πλαισίου και τη μελλοντική μας δουλειά σε σχέση με τις υβριδικές απειλές. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Σύστημα μπορούμε να συμβάλλουμε μαζί με την Εξωτερική Υπηρεσία ώστε να πετύχουμε αυτά αποτελέσματα. Για το EDA. Αν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε τις υβριδικές απειλές θα πρέπει να εστιάσουμε στο capability development, τον κύριο στόχο και έργο της υπηρεσίας μας. Και επ' αυτού και σε σχέση με τον ευρυντικό πόλεμο και απειλές, είχαμε διοργανώσει κάποιες δράσεις για να αντιμετωπίσουμε ακριβώς το τι χρειαζόμαστε σε περίπτωση όπου υπάρχουν αυτές οι απειλές και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Ξεκίνησαμε το Μάρτι φέτος και ευτυχώς μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε πάνω από 80 εμπειρογνώμονες από χώρες μέλη, από την Κομισιόν, από άλλες υπηρεσίες, ε, παρατηρητές του ΝΑΤΟ κλπ. Και ήταν η πρώτη φορά που μια τέτοια ανάλυση επιπτώσεων ευρωτικού πολέμου και ανάπτυξη ικανότητα είχε γίνει, λαμβάνοντα υπόψη την εθνική και την πολυεθνική διάσταση. Τι έμεινε τώρα από αυτή την πρώτη δράση. Καταρχάς, επικεντρωθήκαμε στην φάση εντοπισμού που συμφωνήσαμε όλοι ότι είναι πιο αποφασιστική. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν ένα στρατηγικής ενημέρωσης και δυνατότητα σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο αντίδρασης. Αλλά μια πτυχή αφορά ακριβώς τη δικιά μας την απάντηση. Το πώς οι στρατιωτικές απαντήσεις διαθρώνονται σε σχέση με την απειλή Βέβαια, το πρώτο που έχουμε κατά νου είναι η οργάνωση στρατιωτικής έτσι, ανταπόκρισης. Πρέπει όμως να δούμε και τη λειτουργία της κοινωνίας και την ανταπόκριση όσον αφορά αυτές τις υψηλές απειλές και την δημιουργία αυτής της ανθεκτικότητας. Καταρχάς, ας δούμε τη στρατιωτική απάντηση. Βλέπουμε ότι βασιζόμαστε σε δίκτυα επικοινωνιών και πληροφορικής, όμως και άλλες υποδομές, νερό, ενέργεια κτλ. που και αυτά βρίσκονται σε μια ευάλωτη κατάσταση. Γενικά αναγνωρίσαμε κατά τη διάρκεια αυτής της δράσης ότι τα οπλικά συστήματα θα πρέπει να ενσωματώνονται σε όλη αυτή την επιχείρηση και μελλοντικέ λύσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν πιο υψηλά στάνταρτ, πιο υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά την ανθεκτικότητα σε σχέση με τις ε, προδιαγραφές που είχαμε μέχρι πρόσφατα στον ψυχροπόλεμο. Πρέπει επίσης να εντοπίσουμε τους τομείς όπου θα πρέπει να δράσουμε όσον αφορά τα διάφορα συστήματα, την ε, συλλογή πληροφοριών, αναγνώριση, ιατρικά θέματα, αντικατασκοπία. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν τον Απρίλη στους Υπουργούς Άμυνας. Και το επόμενο βήμα, η επόμενη δράση που ήδη εξάγεται, συνίσταται στο να δούμε το πώς αυτές οι δράσεις μας μπορούν να προχωρήσουν και να φτάσουν στην ουσία αυτής της δυνατότητας που πρέπει να οικοδομήσουμε και πώς θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί ή να αναϊεραρχηθεί. Και νομίζω ότι αυτή η δράση προκάλεσε τον ενδιαφέρον πολλών χωρών, γιατί είδαμε ότι είχαμε συμμετοχή πολλών εμπειρογνωμόνων και χαιρόμαστε πραγματικά που υπάρχει σημαντική υποστήριξη από την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Αυτά από μας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, όλα και πρόεδρος. Ε, ευχαριστώ όλους τους ομιλητές και τους τρεις που μπόρεσαν να συζητήσουν για αυτά τα και να μας διαφωτίσουν για αυτά τα τόσο σοβαρά ζητήματα. Πριν προχωρήσουμε, να σας μεταφέρω ένα δικό μου προσωπικό ερώτημα. Κυβερνοπόλεμος. που αποτελεί ένα από τα εργαλεία του υβριδικού πολέμου. Το γεγονό ότι η ρωσική ομοσπονδία βρίσκεται σε υβριδικό πόλεμο με την Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι αυτό είναι σαφέ πια. Δηλαδή προσπαθούν προσπαθούν λοιπόν να κάνουν κάποια πράγματα που βασίζονται ακριβώς στις πληροφορίες, στην πληροφορική μάλιστα. Και αρκετές φορές είναι επιτυχής. Γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα να ρωτήσω επειδή είναι μια ερώτηση που αφορά περισσότερο την Κομισιόν, να μας πει ο εκπρόσωπός της πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει η Κομισιόν αυτό το μεγάλο ρεύμα αναλυθιών και ψευδών που προέρχονται από τη Μόσχα. Από ό,τι ξέρω το Συμβούλιο πρότεινε στην Κομισιόν να συγκροτήσει μια ομάδα η οποία θα αντιμετωπίσει την παραπληροφόρηση και βλέπω ότι νομίζω ότι έχει συγκροτηθεί μια ομάδα 8-9 ατόμων. Αν όμω το συγκρίνουμε αυτό με τη δύναμη την αντίστοιχη της Ρωσία σήμερα όταν έχουμε να κάνουμε με προμπολισμούς μεγάλου. τότε βλέπουμε ότι η απάντηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι κατάλληλη. Ρωτά λοιπόν η Κομισιόν προτίθεται να ενισχύσει αυτή ακριβώς την ομάδα και το ανθρώπινο δυναμικό με τα καταλα κονδύλια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και Βουρασίς το λόγο τώρα. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Δεν πειράζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρε, εγώ νομίζω ότι γιατί απαντήσατε σε αυτό που ήθελα να πω και εγώ, αλλά τέλο να ξεκινήσω την παρέμβασή μου με μια ρητορική ερώτηση, στην οποία εγώ ίδιος θα δώσω απάντηση. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πόσες φορές συζητήθηκε το θέμα του ευρωπαϊκού πολέμου εδώ στην Επιτροπή Άμυνα στο Κοινοβούλιο. Ήδη το έχουμε συζητήσει δεκάδες φορές αυτό το θέμα και πρέπει να σας πω ότι ήδη έχω μεγάλη γνώση για το πώς εντοπίζει κανείς υβριδικές διανέξεις, ποια χαρακτηριστικά έχει ο υβριδικός πόλεμος. Οπότε σε γενικέ γραμμές μπορούμε να πούμε ότι εδώ στην υποεπιτροπή ήδη έχουμε μπουχτίσει, έχουμε μπουχτίσει με τη συνεχή και αένα ή τέλο πάντων συζήτηση για τον υβριδικό πόλεμο. Και δεν το λέω αυτό ως κριτική για σας, αλλά αφορά ολόκληρη την υποεπιτροπή. Εμείς θα πρέπει να πούμε ότι εντάξει, να δούμε και τι προσδοκίες έχουμε και τι θέματα έχουμε προς συζήτηση, αλλιώς χάνουμε το χρόνο μας εδώ. Αυτό είναι η πρώτη έτσι, παρατήρησή μου. Να πω επίσης ότι επανειλημμένως εδώ στην υποεπιτροπή Αμυνάς έθεσα το θέμα το ότι από τη στιγμή που έχουμε καθορίσει το τι αποτελεί η υβριδική σύγκρουση και διένεξη θα πρέπει να καθορίσουμε ακριβώς και ποια είναι και η απάντησή μας η οποία και από τη φύση και αυτή πρέπει να είναι ευρυδική. Ο ευρυδικός πόλεμος απαιτεί ευρυδικές απαντήσεις. Κάτι το οποίο είναι αρκετά περίπλοκο γιατί σημαίνει ότι διάφορες και πολλές υπηρεσίες πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους. Οπότε τίθεται ένα ζήτημα αποτελεσματικότητας. Οπότε νομίζω ότι εμείς πια δεν έχουμε πιστεί οι ίδιοι ότι είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις υβριδικές απειλές με υβριδικά εργαλεία. Κάθε άλλο πιστεύω ότι εδώ υπάρχουν σοβαρές επικαλύψεις όσον αφορά δραστηριότητες, δράσεις, αναλύσεις κλπ. Και η έννοια ασφάλειας που ακολουθεί ο καθένας η θεωρία υπαρκή, νομίζω ότι τελικά δεν φτάνει. Χθε στην ΑΦΕΤ, στην Επιτροπή ΑΦΕΤ, με τον κύριο Στατίνα, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση από μια Αμερικανική υπηρεσία, η οποία ακριβώς αποδεικνύει την αντίληψη των Ευρωπαίων σε σχέση με τις δράσεις σας, σε σχέση με τα χρήματα που δαπανούνται για αυτές τις δράσεις. Ότι δηλαδή δεν αρκεί σήμερα στην Ευρώπη το να ενισχύσουμε τις ε, δυνατότητες μας. Θα πρέπει να αυξηθούν τα κοντιλία βέβαια για τις ταπάνες που πολλές φορές δεν υπάρχουν βέβαια αλλά δεν υπάρχει έγκριση γι' αυτό το οποίο σημαίνει ότι αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρό πρόβλημα εδώ γιατί εμείς προσπαθούμε να πείσουμε τους πολίτες ότι πρέπει να δαπανίσουμε περισσότερα χρήματα, αλλά πρώτα πρέπει να πείσουμε τους εαυτούς μας. Τώρα, να προχωρήσω στις ερωτήσεις μου, αφού σας έθεσα όλα αυτά. Καταρχάς, σήμερα να ρωτήσω τι δουλειά έχει γίνει ακριβώς ώστε τα ευρωπαϊκά πολιτικά δορυφορικά συστήματα, Κοπέρνικος, Γαλλίο κτλ. να μπορούν να χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς. Έχουν δημιουργηθεί για να προσφέρουν μεταξύ άλλων και μια καλή εναλλακτική σε σχέση με το GPS που είναι αμερικανικό σύστημα. Τι γίνεται με την ασφάλεια στην αεροπλοεία, στις ε, θαλάσσιες μεταφορές, οδικές μεταφορές χρησιμοποιούνται εκεί, αλλά ταυτόχρονα μπορούν να μας επιτρέψουν όλα αυτά να συλλέξουμε πληροφορίες και να προστατευτούμε από πυρηνικές καταστροφές, από οποιοδήποτε άλλα ατυχήματα. Τα συστήματα λοιπόν αυτά, να πούμε όμως ότι ενδιαφέρουν και διάφορες υπηρεσίες κατασκοπίας. Οπότε εδώ θα πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε ώστε να χτίσουμε, να δημιουργήσουμε αυτή την ανθεκτικότητα που λέγαμε. Τώρα, να πω και κάτι άλλο. Στην Ευρώπη υπάρχει πολλή προπαγάνδα, όχι μόνο από τη Ρωσία και από το ISIS. Στο ίντερνετ προσπαθούν να στρατολογήσουν νέους και στο κοινοβούλιο είχαμε ετοιμάσει ένα έγγραφο πρόσφατα για να αντιμετωπίσουμε αυτό τον πόλεμο προπαγάνδας. Να ρωτήσω λοιπόν, εσείς στα οργανά σας, στις υπηρεσίες σας, πώς το αντιμετωπίζετε αυτό, πώς μπορούμε να ενημερώσουμε σωστά τους Ευρωπαίους πολίτες για τις σημαντικές αυτές απειλές που αντιμετωπίζουμε και πώς μπορούμε να αποτρέψουμε αυτές τις ε, πληροφορίες ή πώς τα θεσμικά όργανα της Ένωσης θέλουν να παίξουν ένα ενεργό ρόλο ώστε να αντιμετωπίσουμε ακριβώς αυτή την εκστρατεία παραπληροφόρησης και προπαγάνδας. Πώς να εντοπίζουμε ότι η πληροφορία προέρχεται από αξιόπιστες πηγές και πότε όχι. Τελευταία ερώτηση τώρα για τη χρηματοδότηση. Πώς σας φαίνεται η χρηματοδότηση των πιο σημαντικών ευρωπαϊκών θεσμών σε σχέση με την οικονομική του δυνατότητα να αντιμετωπίζουν τις απειλές που αναφέραμε προηγουμένως, δηλαδή τις απειλές από τον κυβερνό χώρο, επιθέσεις ας πούμε, στις διάφορες ε, εγκαταστάσεις υποδομών, η διείσδυση σε συστήματα πληροφορικής από τη Σκοπιά, απλά και μόνο της άμυνας. Τι άποψη έχετε γι' αυτό, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Στοεύσκη. Μήπω κάποιο άλλο θέλει το λόγο. Μήπως θέλετε να παρατηρήσετε κάτι. Αν όχι, τότε θα ζητήσω από τους συζητητέ μα να απαντήσουν. Νομίζω ότι κυρίω είχαμε δύο ερωτήματα. Ένα από μένα, το πιο απλό, και ένα τριπλό ερώτημα τον κ. Στρουγέσκη. Πριν σας δώσω όμω το λόγο, να ευχαριστήσω τους Πολωνούς και στο Γεύσκι, οι οποίοι σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις βγήκαν πρώτοι οι πιο φιλοευρωπαίοι. 72% είναι ο πιο φιλοευρωπαϊκός λαός στην Ευρώπη. Έχετε το λόγο κύριε, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω να δίνω τις απαντήσεις και στη συνέχεια βέβαια οι συνάδελφοι θα συμπληρώσουν και άλλα στοιχεία. Έχετε δίκιο. Εσείς και τα μέλη της Επιτροπής και εγώ και εμείς που είμαστε εδώ πάνω γνωρίζουμε τι είναι οι υβριδικές απειλές. Αλλά δεν ε, είναι αυτονόητο ότι όλοι γνωρίζουν σε όλα τα κράτη-μέλη τι ακριβώς είναι οι υβριδικές απειλές. Γιατί κάποιες φορές υπάρχουν υποκείμενα που δέχονται υβριδική απειλή και δεν το αντιλαμβάνονται καν. Γι' αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης γύρω από τις υβριδικές απαλληλές γιατί είναι πολύ πιθανό τα υποκείμενα, τα θύματα αυτών των απειλών να μην το αναγνωρίζουν καν. Σημαντικό όμως είναι το γεγονός ότι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρώτη φορά συζητούν τι ακριβώς δράσεις θα αναλάβουν προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υβριδικές απειλές. Και έχουμε για πρώτη φορά ένα έγγραφο το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις και ελπίζουμε να ε, λάβουμε τη συγκατάθεση των ε, κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί είναι πολύ σημαντική η διαδικασία αυτή. Εμείς αντιμετωπίσαμε και το θέμα του αν θα πρέπει να δημοσιεύσουμε μια τέτοια στρατηγική. Γιατί αν δημοσιεύσεις μια τέτοια στρατηγική, αποκαλύπτεις σε έναν βαθμό και τα ευάλωτα σημεία σου. Παρόλα αυτά, ε, εμείς αποφασίσαμε να δημοσιεύσουμε γιατί θεωρήσαμε ότι ήταν η καλύτερη επιλογή για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και ένα τελευταίο σχόλιο. η απάντηση στις υβριδικές απειλές δεν θα δοθεί από ένα μόνο θεσμικό έργανο, την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ή την Επιτροπή. Θα πρέπει να είναι μια κοινή απάντηση και των κρατών μελών, γιατί υπάρχει πιθανότητα να δέχεσαι απειλή ως Τσεχία και ταυτόχρονα η ίδια απειλή να αφορά και την Πολωνία αλλά να μην το συνειδητοποιεί εκείνη η χώρα. Γι' αυτό θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο ότι το πραγματικό ζητούμενο είναι η συνεργασία. Για το διάστημα και το συγκεκριμένο ερώτημα που θέσατε για τον Γαλιλαίο. Εμείς εξετάζουμε την εκπόνηση μιας στρατηγικής για το διάστημα έως το τέλος της φετινής χρονιάς που θα λαμβάνει υπόψη και θα εξετάζει την πιθανότητα αξιοποίησης του διαστήματος στο μέλλον. Για τον Γαλιλαίο. Το Γαλιλαίο είναι ένα πρόγραμμα μη στρατιωτικού χαρακτήρα. χαρακτήρα. Σε αντίθεση με το, το GPS, το οποίο ήταν αρχικός στρατιωτικό πρόγραμμα. Βεβαίως, οι υπηρεσίε που παρέχει το Γαλιλαίο, ε, ε, στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνεται και το PMS, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τον Γαλιλαίο και για ανταλλαγή μυστικών πληροφοριών. Πολλά κράτη-μέλη είναι πρόθυμα να χρησιμοποιήσουν και να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα μόλις ε, ολοκληρωθεί και τεθεί στη διάθεσή μας. Το Γαλιλαίο λοιπόν μπορεί να αποτελήσει ένα από τα στοιχεία της απάντησης που θα δώσουμε. Όσον αφορά το Κοπέρνικους, είπατε σωστά είναι ένα εργαλείο παρακολούθησης και παρατήρησης. Εμείς πραγματικά πιστεύουμε και εξετάζουμε ποιες δυνατότητες έχουμε για να αξιοποιήσουμε το Κοπέρνικους για ε, λόγους ασφάλειας. Φυσικά όλα αυτά μπορούν να συνδυαστούν και με άλλα ζητήματα όπως τα μη επανδρομένα αεροσκάφη κτλ. Αλλά πιστεύουμε ότι όλοι οι δορυφόροι που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και για την ασφάλεια. Εδώ ε, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και να, να συνυπολογίσουμε και το θέμα της, μετανές, της μετανάστευσης. Για το δεύτερο ερώτημά σας που συνδέεται σε ένα βαθμό με αυτό που είπατε για τις κυβερνοεπιθέσεις που δεχόμαστε και τις σχετικές απειλές. Όπως είπα, η απάντηση θα πρέπει να είναι συλλογική. Το θέμα δεν είναι μόνο να εξευρεθούν οι πόροι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα είναι να υπάρξει συνεργασία. Αναφερθήκατε στη Ρωσία στο Ισλαμικό κράτος θα μπορούσε να είναι και κάποιος άλλος. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαίο να υπάρξει μια συλλογική απάντηση και να χρησιμοποιηθούν από κοινού όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήνυμα όμως που στέλνει και η ανακοίνωση είναι ότι θα πρέπει τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας να ενισχυθούν και η ευαισθητοποίηση και η πολιτική συζήτηση που θα ακολουθήσει στα κράτη-μέλη ε, θα βοηθήσει ακριβώς σε αυτό το πράγμα. Να ε, ενισχυθούν οι πόροι, γιατί σε κάποια κράτη-μέλη η αναγκαιότητα είναι σαφής, σε κάποια άλλα κράτη-μέλη ε, η αναγκαιότητα αυτή δεν έχει γίνει ακόμα πλήρως κατανοητή. Για την κυβερνοασφάλεια. Φυσικά πρόκειται για πολύ σημαντικό στοιχείο προστασίας. Γνωρίζετε ότι εργαζόμαστε πάνω σε αυτό το θέμα ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει σχεδόν έτοιμη και μια οδηγία. Θα πρέπει ακόμη να εγκριθεί και να εφαρμοστεί βεβαίως. Αλλά υπάρχει συμφωνία από τα κράτη-μέλη. Αλλά εκεί στην πρόταση αυτή αναδεικνύεται ότι χρειαζόμαστε καλύτερους μηχανισμούς για να αποκρούσουμε στο μέλλον πιθανές κυβερνοεπιθέσεις. Για τη ριζοσπαστικοποίηση και τη χρήση του διαδικτύου για, ριζοσπαστικοποίηση, για σκοπούς ριζοσπαστικοποίησης, εμείς στην Κομισιόν εξετάζουμε τι μπορεί να κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί θέλουμε να συνεργαστούμε και με διάφορους ενδιάμεσους, με την Google και άλλες εταιρείες, προκειμένου αυτού του είδους το περιεχόμενο να μην διατίθεται σε νέους ανθρώπους αλλά και ευρύτερα στο κοινό. Είναι ένα από τα μέτρα που εμείς θέλουμε να εφαρμόσουμε, να αναγκάσουμε ή εν πάση περιπτώσει να παρατρύνουμε τους ενδιάμεσους να μην φιλοξενούν τέτοιου είδους ε, περιεχόμενο που οδηγεί στη ριζοσπαστικοποίηση. Να δώσω το λόγο στον συνάδελφο. Ευχαριστώ πολύ, ήταν πολύ πλήρη η απάντησή σας. Να πω όμως και εγώ ορισμένα πράγματα. Η κοινή ανακοίνωση και η όλη προσπάθεια αφορά το να βρούμε ποια είναι η βοήθεια που μπορεί να παράσχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν αυτά τις υβριδικές απειλές. Πρόκειται για εθνική αρμοδιότητα. Κανείς δεν πρόκειται να παρέμβει στα εσωτερικά των κρατών μελών. Τα ίδια τα κράτη-μέλη πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αλλά εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε. Ενδεχομένως να υπάρχουν τομεί όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να παρέχει ε, σημαντικότατη υποστήριξη και βοήθεια. Προκειμένου ένα κράτο μέλο να μπορεί, για παράδειγμα, να σχηματίσει μια συνολικότερη εικόνα για το τι συμβαίνει. Μπορεί να λαμβάνει πληροφορίε πρώτα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για την αναθεκτικότητά του. Και όπω υπόθηκε, υπάρχει ήδη ε, μια οδηγία ε, η οποία προβλέπει την, ε, την συνεργασία σε ζητήματα κυβερνοχώρου. Και είναι κρίσιμη σημασία γιατί στον κλάδο υπάρχουν ήδη συγκριτικοί δείκτες προκειμένου να υπάρξει ευαισθητοποίηση γύρω από τα ελάχιστα κριτήρια που ισχύουν και αυτό αποτελεί προσπάθεια της Κομισιόν. Είναι η ρυθμιστική ε, αρμοδιότητα ακριβώς λόγω της, του γεγονότος ότι είμαστε διασυνδεδεμένοι. Κανείς δεν μπορεί να σηκώσει τείχου γύρω από τη χώρα του και να πει ότι εγώ μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Δεν γίνεται αυτό. Είμαστε διασυνδεδεμένοι και αλληλοεξαρτώμενοι. Επικοινωνίες. Το βλέπουμε εκεί. Πρέπει, χρειαζόμαστε ενότητα. Έχουμε δει ποιες είναι οι επιπτώσεις όταν αφήνουμε τους αντιπάλους μας να μας διχάζουν και να μας διαιρούν. Αντιθέτως, ισχύσεν τη ενώση. Αλλιώς, είμαστε ευάλωτοι. Αλληλεγγύη. Είναι κρίσιμο θέμα η αλληλεγγύη. Αποτελεί τη συγκολητική ουσία που μπορεί να παράσχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαδικασία αυτή, προκειμένου να την ενασχίσει. Και οι ευρυδικές απειλές αποτελούν ένα έδαφος όπου πραγματικά είναι απαραίτητο η ευρωπαϊκή κοινότητα να εκφράζει και να εφαρμόζει την αλληλεγγύη της στην πράξη. Ο κυβερνοχώρος προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες, το γνωρίζουμε όλοι, αλλά προσφέρει και τις δυνατότητες σε εκείνους που το θέλουν να προκαλέσουν κακό. υπάρχουν και σχετικές εκτιμήσεις που λένε ότι οι οικονομικές απώλειες που οφείλονται σε κυβερνοπεθέσεις κατ' έτος, σε ολόκληρο τον χρόνο, ανέρχονται σε ένα τρισεκατομμύριο ευρώ. Είναι πάντως σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι και οι κυβερνοεπιθέσεις αποτελούν σημαντικότατο τμήμα του τρόπου με τον οποίο διεξάγονται οι πόλεμοι στη σύγχρονη εποχή. Και θα πρέπει και εμείς να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε τον κυβερνοχώρο, αν παρουσιαστεί η ανάγκη. Άλλο συμπέρασμα, και γι' αυτό η Κομισιόν, είναι, ε, και η Κομισιόν θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό παράγοντας. Πρέπει να συνεργαστούμε με τις επιχειρήσεις. Ο κυβερνοχώρος δεν αφορά μόνο τις κυβερνήσεις. Χρειάζεται η συνεργασία και με τις μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ίντερνετ. Αυτά, αυτές είναι που διαμορφώνουν το μέλλον μας, που διαμορφώνουν τα δίκτυα που εμείς χρησιμοποιούμε. Και για να μπορούν οι κυβερνήσεις να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις σήμερα για αύριο, χρειάζεται ως απαραίτητος όρος η συνεργασία με αυτές τις εταιρείες. Πολλές ερωτήσεις αφορούσαν το, θέμα της προπαγάνδας. Η απάντηση δεν είναι αντιπροπαγάνδα. Το να απαντήσεις σε έναν κεντρικό μηχανισμό προπαγάνδας. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν άλλον μηχανισμό, να δημιουργήσουμε έναν άλλον μηχανισμό για να κάνουμε αντιπροπαγάνδα. Εμάς το όπλο μας είναι η ενημέρωση. Για το πώς χρηματοδοτούνται διάφορες έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις. Θα υπάρξουν στο μέλλον συζητήσεις για το πώς μπορούμε να μειώσουμε την ευαλωτότητά μας στο μέλλον. Η εκπαίδευση, η παιδεία είναι πάρα πολύ στο τομέας. Πώς θα προλάβουμε αυτήν την προσπάθεια μαζικής πλήσης εγκεφάλου την οποία κάνουν διάφορες τρομοκρατικές οργανώσεις. Αυτά. Uh, ευχαριστώ. Νομίζω ότι τα περισσότερα υπόθηκαν. Από τη σκοπιά της ΑΓΕΤ να τονίσω το εξή. Όπως είπε και ο Πιέρ, βρισκόμαστε στην αρχή Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Αλλά να κατανοήσουμε ότι ήδη έχουμε προχωρήσει πολύ. Γιατί είναι η πρώτη φορά που κάνουμε κάτι μαζί. Η ΕΕΔ, η Κομισιόν, διάφορα οργανισμοί συνεργάστηκαν. Εδώ ο μόνος φοβός είναι οι χώρες μέλη και σε αυτές στρέφομαι. Και οι χώρες μέλη πρέπει να δράσουν σωστά ώστε να μην έχει αδύναμους κρίκους η αλυσίδα. Θα πρέπει να κατανοήσουν οι χώρες μέλη, θα πρέπει να συνεχίσουν να διαθέτουν κονδύλια και να μοιράζονται πληροφορίες ώστε να γίνουμε πιο ανθεκτικοί. Γιατί προς την ανθεκτικότητα την όλες μας οι προσπάθειες και μετά από αυτά που δημιουργήσαμε μέχρι τώρα μπορούμε να πάμε μετά στην επόμενη φάση όπου θα λέμε ναι, Έχουμε τον έλεγχο, αν όχι πλήρω, αλλά τα περισσότερα τουλάχιστον τα ελέγχουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος. Ακούσαμε μια έτσι σχεδόν ανώνυμη κλίση, κάλεσμα για Ευρωπαϊκή Ενότητα, λέει ο Πρόεδρος. Το οποίο θα μας ε, κάνει να είμαστε έτσι νικητές στο πεδίο της ενημέρωσης. Να δούμε λοιπόν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Κύριε Στρέφη, ναι. θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ναι. Έχουμε χρόνο, οπότε θα υποφεληθώ. Να πω ότι η κατάσταση είναι κάπως ιδιαίτερη. Γιατί βλέπω ότι δεν είναι εδώ κανένα ευρωβουλευτή. Υπάρχουν πιο πολλοί εισηγητέ και αποσιάζουν όλοι οι βουλευτέ. Πάντω ευχαριστώ για αυτά που είπατε. Βλέπω ότι συνειδητοποιούμε τις, τι δυσκολίε υπάρχουν. Βέβαια θα μπορούσε να πει κανεί ότι δεν είμαστε και τόσο σοβαροί, επειδή λέμε ότι εντάξει, η αλληλεγγύη είναι πολύ σοβαρό θέμα, τη στιγμή που κοντεύουμε να έχουμε και Brexit σε λίγο. Οπότε, τι γίνεται όταν ένας αδύναμος κρίκος καθορίζει τη δύναμη όλης της αλυσίδας. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ευρώπης κιόλας, γιατί έχουμε πολλούς και διάφορους αδύναμους κρίκους και δεν θέλω να κατονομάσω κανένα. Αλλά τέλο πάντων, να αποφεληθώ σε ευκαιρία για να σας δώσω κάποιες πληροφορίες. Η συζήτηση που αναφέραμε προηγουμένω για τα δορυφορικά συστήματα, Κοπέρνικος και Γαλιλαίος. Εκεί είδαμε τις διάφορε θέσει και στάσεις που υπάρχουν στο Κοινοβούλιο και είδαμε να υπάρχουν και αντικρουόμενε προσδοκίε για αυτό το θέμα. Οι πράσινοι α πούμε θέλανε ο Κοπέρνικος να χρησιμοποιείται μόνο για την αναζήτηση πεταλούδων και λουλουδιών. και είχαν προσθέσει πράγματα που δεν αφορούσαν μόνο την πτυχή της άμυνας. Άλλοι πάλι από την αριστερά έλεγαν ότι εντάξει στην αρχή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Κοπέρνικο για τους ε, πρόσφυγες άλλαξαν με τα γνώμη, στην αρχή ήταν θετική γιατί ενσύγησαν ότι μπορούμε έτσι να χρησιμοποιούμε τα συστήματα αυτά για την επιστροφή των προσφύγων. Οπότε βλέπετε ότι υπάρχουν πολλές φορές αντιφάσεις. Μετά να προχωρήσω. Αναφερθήκατε στα μη πανδρομένα. Σήμερα υπάρχει τεράστιος αριθμός τους στην Ευρώπη. Υπάρχουν μη έδρομενα σκάφη τα οποία μεταφέρουν πολύ σημαντικά χημικά για την καταπολέμηση των ζυζανίων στην Γεωργία και πετάνε σε ύψος 1200-1500 μέτρα. Οπότε το ερώτημα είναι κατά πόσο οι χώρες μέλη μπορούν να αποδεχτούν νομοθεσία ώστε αυτά τα μη επανδρομένα σκάφη να μην χρησιμοποιούνται από τρομοκράτες. Μέχρι στιγμής έχουμε κανόνες για τα στρατιωτικά σκάφη αυτού του είδους. Αν όμως ανακύψουν άλλα προβλήματα, τότε οι χώρε πρέπει να κάνουν και αυτές υποχωρήσει. Και δυστυχώς ο πιο κοινό παρονομαστής σε επίπεδο οδηγία πρέπει να είναι βέβαια αντικείμενο συνένεσης πανευρωπαϊκής. Πρέπει να υπάρχει μια συνοχή. Οπότε εγώ αυτό που βλέπω να λείπει είναι μια δυνατότητα ταχεία ανταπόκρισης όσον αφορά τις απειλές οι οποίες προέρχονται εκτός Ευρώπης. Εμείς χαιρόμαστε που ερχόμαστε σε συναντήσεις και συζητήσεις όπως η σημερινή ώστε να έχουμε τέλο πάντων μια κοινή αντίληψη για τι απειλέ. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλέ εκεί έξω, αλλά για την ανταπόκριση στι απειλέ είμαστε σχετικά αργοί. Και υπάρχει και μια ερώτηση που δεν απαντήσατε για τα κονδύλια, για τη χρηματοδότηση, τα αιτήματα χρηματοδότηση. Τι γίνεται. Πάντως, ε, να σας ευχαριστήσω όλους τους ηγητές που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας, γιατί είναι σημαντικό να μαθαίνουμε περισσότερα και να προετοιμαζόμαστε καλύτερα εδώ στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, για το θέμα της αλληλεγγύης. Σε μια εβδομάδα λέτε μπορεί να έχουμε και Brexit. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ελπίζω να μην συμβεί αυτό, να δούμε το αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, να πω εγώ ότι ναι, έχουμε δυσκολίες, αλλά ποια είναι η εναλλακτική. Αν δεν υπάρχει αλληλεγγύη θα χάσουμε όλοι. Δεν υπάρχει λοιπόν άλλη επιλογή. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να υπάρχει αλληλεγγύη. Μπορεί να μην είναι βέβαια πάντοτε αποτελεσματική, μπορεί να υπάρχουν και κλπ. Αλλά τι είναι εναλλακτική, τι άλλη λύση έχουμε. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να παλεύουμε, γιατί αν δεν υπάρχει αλληλογή δεν θα λειτουργήσει τίποτα. Για το διάστημα τώρα και τη χρήση του Γαλιλαίου, του Κοπέρνικου, αυτών των συστημάτων. Να είμαστε ξεκάθαροι. Αυτά τα συστήματα θέλουν να κάνουν κάποια πράγματα. Έτσι, εντάξει το να παρακολουθούν ας πούμε, λουλούδια, εντάξει, αλλά και άλλα όπως παρακολούθηση του επίπεδου των ρήπων, της ροής των μεταναστών κτλ. κτλ. Υπάρχει όμως ένα κόστος, έτσι. Το θέμα είναι θα στείλουμε ένα δορυφόρο για τους δρύπους, έναν άλλο για τους ε, μετανάστες, έναν άλλο, μετα... έναν άλλο συγγνώμη, δορυφόρο για να παρακολουθεί κάτι άλλο. Υπάρχει μια τιμή, ένα τίμημα που πρέπει να πληρωθεί. Έτσι. Και αυτό αφορά τις χώρες μέλη. Και βέβαια αφορά το Κοινοβούλιο και την χώρα μέλος να αποφασίσει το τι θέλει να πληρώσει και τι προτεραιότητες έχει στα πλαίσια του προπολογισμού της Ένωσης. Υπάρχει κόστος λοιπόν, αλλά πρέπει να αναλυθεί και πρέπει το Κοινοβούλιο να θέσει προτεραιότητες μετά από συμφωνία με τις χώρε μέλη για τη μελλοντική χρήση του Κοπέρνικου και των άλλων παρόμοιων συστημάτων. Για τα μη επανδρομένα. Δεν έχουμε πανευρωπαϊκή νομοθεσία. Έχουμε σε κάποιες χώρες, αλλά όχι σε όλες. Είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε. Περίπλοκο είναι όμω, γιατί πρέπει να δούμε τι γίνεται με την αεροπλοεία, ώστε να βρούμε μια ισορροπία δεν είναι εύκολο, αλλά συμφωνώ με την διάδοση των σκαφών αυτών επιβάλλεται να βρούμε μια λύση. Τέλος, χρηματοδότηση. Επαρκεί, μάλλον όχι, αν θέλετε να το πούμε απλά. Ξέρουμε όμως ότι πρέπει να δράσουμε στο υπάρχον νομοθε... Συγγνώμη, δημοσιονομικό πλαίσιο, οπότε πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Στο μέσο μέλλον θα έχουμε την έκδοση κανόνων και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει ποιες είναι οι προτεραιότητες μας εδώ. Δεν λέω ότι εσείς δεν και καλά πρέπει να αποφασίσετε τώρα, αλλά θα πρέπει να δείτε συνεργασία με τις χώρες ποιο θα μπορούσε να είναι το καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα. περάμε στις Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους πήραν μέρος σε αυτό το πάνελ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό, να ευχαριστήσω και όλους σας που ήρθατε, που πήρατε μέρος στη σημερινή συνάντηση. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους διερμηνείς για την εργασία τους. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε αύριο στις 9 την ίδια αίθουσα. Καλό σας βράδυ.